Busy, huh? You had another minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti, ambasciatori. Καλώς, ε, καλώς ήρθατε. Κύριε Πρέσβη, τα σέβη μας. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον Σάντορ Φατσέκας, ε, Ούγγρο Υπουργό Γεωργίας και Ανάπτυξης, ε, προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Να καλωσορίσουμε επίσης ε, και τον Υπουργό και τον Πρόεδρο Σαντόρ. Κύριε, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα για να μας πείτε τις εξελίξεις για το μέλλον της Γεωργίας σε συνέχεια της συζήτηση που κάνατε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την έκθεση του Albert Des, μια έκθεση που θέλει να απαντήσει στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18 Νοεμβρίου του 2010 και καθώς επίσης και να καθορίσουμε και τις προτεραιότητες που εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας ε, θεωρούμε πιο σημαντικές. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα και σας δίνω απευθεία το λόγο. Παρακαλώ.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 μου ζήσατε να επιστρέψω, να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις εργασίες του Συμβουλίου, προετοιμάζοντας το μέλλον της ΚΑΠ. Και γι' αυτό ανέλαβα την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα, υπό, ε, προεδρικής, υπό Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε δραστηριότητες επίπεδου προεδρίας που να είναι σε συνεργασία πάντα με το Κοινοβούλιο. Και σε αυτό το κλίμα βαρευρίσκομαι εδώ, ενώπιόν σας και χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου σε, με μεγάλη πλειοψηφία τις, ενέκρινε τις προτεραιότητες της ε, Ουγγρικής Προεδρίας δίνοντας ε, τις ε, τους προσανατολισμούς για την, το μέλλον της ΚΑΠ. Ανάμεσα στα θέματα τα γεωργικά. Η, Ουγγρική Προεδρία έδωσε προτεραιότητα στις ε, διαπραγματεύσεις για την ε, επικοινωνία με την ε, Επιτροπή, καθορίζοντας το μέλλον της ΚΑΠ, γνωρίζοντας ότι η γεωργία αποτελεί έναν στρατηγικό τομέα της Ευρώπης, μια σημαντική αξία της Ευρώπης και της οικονομικής ανάπτυξής Από την αρχή η Ουγγρική Προεδρία εξέφρασε την φιλοδοξία της να ε, λάβει να εξασφαλίσει όσο μεγαλύτερη σύγκληση για την ΚΑΠ μέχρι το 2020. Και έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι όταν ε, τις 17 Μαρτίου το 2011 το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα της Προεδρίας για το μέλλον της ΚΑΠ με ενισχυμένη πλειοψηφία. 20 μέλη ήταν υπέρ. Η ενισχυμένη πλειοψηφία είναι ένα σημαντικό ε, μήνυμα για την ε, ενίσχυση της ΚΑΠ. Ε, είναι ένα καλό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες, τους αγρότες και προς όλους αυτούς που ζουν στις αγροτικές περιοχές, όλους τους ενδιαφερομένους από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ. Πιστεύω ότι μέσα από τα συμπεράσματα της ε, Προεδρίας έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ε, πρέπει να υπογραμμίσω ε, ότι βρήκαμε ένα κοινό παρονομαστή. Βέβαια, υπάρχει, πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσο διαφορετικά είναι τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό προς ε, το καλό όχι μόνο των ε, Ευρωπαίων γεωργών αλλά και για το καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Τα συμπεράσματα εκφράζουν με σαφήνεια την θέση της ενισχυμένης πλειοψηφία των κρατών μελών και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα συμπεράσματα έδωσαν τους απαραίτητους προσανατολισμούς προς την Κομισιόν για να κάνει τις δικές της νομοθετικές προτάσεις ε, στηριζόμενοι στις αρχές που εκφράστηκαν στην ανακοίνωσή της. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να συνοψίσω με συντομία την ουσία των συμπερασμάτων της Προεδρίας. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τους τρεις στόχους για το μέλλον της ΚΑΠ όπως διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Η Ευρώπη θα πρέπει να παράγει αρκετά ε, τρόφιμα, επαρκή τρόφιμα, ε, ασφαλή και με καλή ποιότητα και ε, σε προσιτές τιμές. Θα πρέπει να γίνει ευφύς διαχείριση των φυσικών μας πόρων, σεβασμός προς το περιβάλλον, το κλίμα, την ευζοία των ζώων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και μια ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας τους να παραμείνουν οικονομικά αηφόρες και βιώσιμες. Ανάμεσα στα συμπεράσματα θα τόνιζα το γεγονός ότι οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πεπισμένοι ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ένας ε, αηφόρος γεωργικός τομέας, παραγωγικός και ανταγωνιστικός, θα οδηγήσει σε μια σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική ε, θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή στο μέλλον και θα πρέπει να έχει ε, ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους που να είναι αναλογικοί προς τους, τα, ε, τους σκοπούς της. Οι προτάσεις ε, δέχονται ότι το χρηματοδοτικό πακέτο βέβαια θα καθοριστεί από το Συμβούλιο. Η δομή, η τρέχουσα δομή της ΚΑΠ στηριζόμενη σε δύο σαφείς και συμπληρωματικούς πυλώνες πρέπει να διατηρηθεί. Η απλούστευση της ΚΑΠ, ένα από τα πιο ακαθόδια ερωτήματα. Το Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να εξετάσει τις προτάσεις που έκαναν τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο αυτό. Τα συμπεράσματα αναγνωρίζουν την ομιμότητα των άμεσων πληρωμών που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των αγροτών. Τους τελευταίους μήνες διεξάγεται ένας έντονος διάλογος για την ανακατανομή των αμέσων πληρωμών στα εισοδήματα των γεωργών. Στα συμπεράσματα βλέπουμε ότι στο μέλλον αυτή η ανακατανομή πρέπει να γίνεται πιο ισότιμα, αλλά το γενικό πλαίσιο του προϋπολογισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη φυσικά και κάθε σημαντική αλλαγή που θα μπορούσε να προκαλέσει στευλώσεις θα πρέπει να αποφεύγεται. Το Συμβούλιο είναι ε, ανοιχτό ε, σε πιο στοχοθετημένες ε, ενισχύσεις γιατί έτσι θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια. Ταυτόχρονα έχουμε δει μια μεγάλη αντίσταση στην ιδέα της οριοθέτησης των ε, ενισχύσεων που δίνονται σε ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Το Συμβούλιο φυστά ε, την προσοχή της Κομισιόν στο γεγονός ότι αν επιθυμεί να ε, κάνει μια πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να την κάνει χωρίς να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και την απλούστευση της ΚΑΠ. Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα πρέπει να ε, παραμένει ε, στοχευμένη στην αγορά και ανταγωνιστική. Οι Υπουργοί της Ένωσης θεωρούν ότι είναι σημαντικό η γεωργία να παραμείνει αηφόρος, βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική. Τα κράτη-μέλη επιθυμούν να θέσουν τέρμα στην μείωση των εσόδων των γεωργών. Το Συμβούλιο έχει καταδείξει την δέσμευσή του στην προστασία των γεωργών από τους αυξανόμενους κινδύνους που ε, προκαλούνται από τις ε, διακυμάνσεις των τιμών και των εσόδων. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν μέτρα αγοράς ως ε, δικλείδα ασφαλείας. Τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν επίσης την ιδέα ότι η παραγωγή θα μπορούσαν να έχουν ισότιμη ε, συμμετοχή στα έσοδα της διατροφικής αλυσίδας. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους επίσης. Υπάρχει συνένεση στο πρασίνισμα το λεγόμενο της ΚΑΠ και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν επίσης ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να ανταποκριθεί και στις κλιματικές αλλαγές. Αυτό το πρασίνισμα θα πρέπει να είναι μια, σε συμφωνία με τους στόχους της απλούστευσης της ΚΑΠ. Α, λοιπόν, δεν μπορούν να αυξήσουν τη, τα έξοδα των γεωργών, τα διοικητικά ή των διοικήσεων των κρατών μελών το πρασίνισμα θα πρέπει να λάβει υπόψη ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των γεωργών και της κοινωνίας, αλλά και τις πραγματικότητες της οικονομικές που ισχύουν. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, ε, στους στόχους τους περιβαλλοντικούς και τους γεωργικούς παρά μόνο με την βοήθεια της καινοτομίας. Η ΚΑΠ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα εφαρμόσει τα αποτελέσματά της. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΚΑΠ έχει αποδείξει την νομιμότητά της. Μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ισχυρή και ευέλικτη παραμένει καθοριστική στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον εξυγχρονισμό και την αηφορία της γεωργίας. δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους νέους γεωργούς. Εναπόκειται σε αυτούς να εξασφαλίσουν την ε, παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη σε επαρκείς ποσότητες, ε, με ασφάλεια και καλή ποιότητα. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή και η συνέργεια ανάμεσα στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις άλλες πολιτικές της Ευρώπης που είναι συναφείς. Και επίσης έχουμε δεσμευτεί να διατηρήσει η Ευρώπη την ποικιλότητα της αγροτικής δραστηριότητας και να βελτιώσει τις ευκαιρίες της οικονομικές των αγροτικών περιφερειών. Σήμερα δεν έχω πρόθεση να σας δώσω ένα πλήρ κατάλογο των συμπερασμάτων, γιατί φυσικά μπορείτε να τα δείτε στα δημοσιευμένα έγγραφα. Ταυτόχρονα υπογραμμίζοντας αυτά τα πιο σημαντικά σημεία, ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το Συμβούλιο έχει δώσει ε, σαφείς προσανατολισμούς και συνεκτικούς σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ και έχει δεσμευτεί έτσι ώστε μια ισχυρή ΚΑΠ να ανταποκριθεί στους στόχους μιας ισχυρής Ευρώπης μέχρι το 2020. Δίνουμε ε, μεγάλη σημασία στις εργασίες του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η έκθεση του κ. Ντες έλαβε πάνω από 1.200 τροπολογίες. Θα είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να καθορίσει συνεκτικούς προσανατολισμούς που να υποστηρίζουν επίσης μια ισχυρή ΚΑΠ. Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας πληροφορήσω επίσης ε, για τα άλλα ε, νομοθετικά ντοσιέ τα οποία θεωρούμε ως προτεραιότητα υπό Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα να τονίσω το πακέτο που αφορά το γάλα και την πολιτική ποιότητας οι γεωργοί και οι καταναλωτές επιθυμούν αυτά να εγκριθούν. Και είναι δική μας κοινή πολιτική ευθύνη να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, εάν είναι δυνατόν, στα πλαίσια της Ουγγρικής Προεδρίας. Επίσης, έχουμε επιτελέσει μεγάλες προόδους εντός του Συμβουλίου σχετικά με την ρύθμιση ε, στην ε, την βασική ρυθμίση της ΚΑΠ. Ε, ε, έχουμε πάνω από χίλιες σελίδες νομοθετικών πράξεων αυτή τη στιγμή και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί αυτή την, την, την διαδικασία επίσης ως προτεραιότητα και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ε, τριμερείς διαβουλεύσεις πρώτης ανάγνωσης. Ανάμεσα στα θέματα τα ρύθμισης, αναμένουμε μεγάλες προόδους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και των αμέσων πληρωμών. Θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω για την, τον ίδιο δυναμισμό που έχει η Ουγγρική Προεδρία ε, στο δεύτερο εξάμεινο. Είμαστε πάντα έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας στις διαβουλεύσεις και για να επιτευχθεί η απαραίτητη πρόοδο στηρίζομαι επίση στη δική σα συνεργασία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε Υπουργέ Φαζέκα. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε σημείο σύγκληση με την Ουγγρική Προεδρία, ώστε το πακέτο γάλα, το πακέτο ποιότητα, τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και των άμεσων πληρωμών να διευθετηθούν. Πολλά ψηφίσαμε, από αυτά τα ψηφίσαμε ήδη στην ε, ε, Επιτροπή μας και ελπίζουμε να έχουν αίσιο τέλος. Βέβαια ελπίζουμε ότι και από πλευρά Συμβουλίου θα υπάρξει αποδοχή των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει σημείο συνεννόησης. Να ξεκινήσουμε τώρα τη γενική συζήτηση. Θα δώσω απευθεία το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, ε, Υπουργό Φατζέκας που βρέθηκε εδώ σήμερα για να μας παρουσιάσει την ε, θέση της Ουγγρικής Προεδρίας και του Συμβουλίου. Με μεγάλη προσοχή άκουσα αυτά που μας αναφέρατε σήμερα. Πολλά εξ αυτών μπορούμε να τα τονίσουμε. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τους στόχους, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε ότι θα συνεχίσουμε να φροντίσουμε για την υψηλή ποιότητα των τροφίμων στην Ευρώπη. Αυτό χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να φροντίσουμε για την προστασία των ζώων, την ενίσχυση της υπαίθρου, όχι μόνο για να επιβιώσει, αλλά για να ενισχύσει πραγματικά. Και για την ε, αηφόρο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία που χρειαζόμαστε. Δικαίως αναφέρατε ότι το καθαριστικό ζήτημα στο τέλος των διαβουλεύσεων είναι το πόσα χρήματα θα διατεθούν στο μέλλον στην αγροτική πολιτική. Μόνο εφόσον έχει απαντηθεί το ερώτημα αυτό, θα μπορέσουμε να λάβουμε οριστικέ αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική η αγροτική του μέλλοντος. Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί σας και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ότι χρειαζόμαστε και τους δύο πυλώνες. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν οι δύο πυλώνες. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς προκειμένου να είναι όσο πιο ευρεία γίνεται η υποστήριξη της διαμόρφωσης τους δύο πυλώνες. Το ένα δύσκολο θέμα και σε εμά αλλά και στο Συμβούλιο και θα πρέπει να αποφασιστεί είναι η κατανομή των ε, δημοσιονομικών πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Και πολλές από τις τροπολογίες αναφέρονται σε τέτοια συντήματα Φυσικά, εδώ ανάλογα με τα συμφέροντα διαφέρουν και οι απόψεις και μάλιστα κατά πολύ. Αλλά σε τελική ανάλυση νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ε, μέσων στην Ευρώπη. Μιλήσατε για τα ανώτατα όρια. Μας το συζήτησε μάλλον και η Γερμανίδα υπουργό ε, Γεωργίας. Στους συντονιστές ήρθε και είπε ότι είναι δύσκολο να βρούμε ρύθμιση χωρίς γραφειοκρατικό άχθος. Και αν δεν έχει νόημα να επιβάλλουμε ανώτατα όρια χωρίς έλεγχο. Νομίζω ότι μεταξύ Κοινοβουλίου και μεταξύ Συμβουλίου υπάρχει η συμφωνία ότι θέλουμε μια γεωργία προσανατολισμένη στην αγορά, όχι όμως ε, ε, μια γεωργία η οποία θα είναι ελεύθερη, θα είναι θύμα της ε, γεωργίας, της, συγγνώμη, της αγοράς. να μην επαφείτε δηλαδή στις μεγάλες διακυμάνσεις ε, που πλήττουν και την γεωργική αγορά. Χαίρομαι που θίξατε και το θέμα των νέων γεωργών. Διεξάγουμε συζητήσεις και με τους νέους γεωργούς και διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις για τον προσανατολισμό της ε, πολιτικής γεωργίας ε, είναι διαφορετικές, πολύ διαφορετικές. Θα ήθελα γενικά να σας ευχαριστήσω, Υπουργέ Βαζέκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Ελπίζω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις σας στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον Αλμπερντές, ο Λουίς Καπουλασάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη αλλά Νομίζω ότι βάσει το την οργάνωση εργασίας ε, η... αυτό σημαίνει ότι η παρουσίαση της, ε, ε, του Υπουργού είναι στο σημείο 13. Έτσι είναι. Σωστά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς τον Υπουργό για την ενημέρωση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, συμπεράσματα τα οποία ικανοποιούν τους σοσιαλιστές διότι υπάρχουν αρκετά σημεία σύγκλησης στα θέματα που μας απασχολούν. Βεβαίω για τα νότατα όρια δεν συμφωνούμε, αλλά εξ των σοσιαλιστών θα ήθελα να πούμε ότι από τις 1267 τροπολογίες που παρουσιάστηκαν, η ομάδα των σοσιαλιστών έκανε τεράστια προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει όσο το δυνατόν τις ε, προτάσεις για τροπολογίες που έκανε λιγότερο από το 10% των τροπολογιών είναι τροπολογίες σοσιαλιστών. Το 10% όμως αυτό το 100% έχει προκύψει από πολύ σημαντική συνένεση μεταξύ όλων των μελών της ομάδας των σοσιαλιστών. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να δείξουμε ότι υπάρχει μεγάλη συνοχή στις προτάσεις που κάνουμε ως πολιτική ομάδα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ ε, σε αυτά που θα πει ο Στέφανο ούτως ή άλλως ο σκιώδης εισηγητής για την άποψη της πολιτικής μας ομάδας αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι η πολιτική μας ομάδα ενδιαφέρεται για αυτό το συμβιβασμό, ένα συμβιβασμό ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη συνοχή της στρατηγικής που παρουσιάζεται. Ευχαριστώ, κύριος Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας και την παρουσίασή σας την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια τροφίμων, να υπάρχει συνένεση για το πρασίνισμα της γεωργίας. Ε, μπορεί βέβαια να υπάρχει συνέντευξη από αυτού, αλλά δεν είμαστε σαφείς ως προς την άγουσα που θέλουμε να ακολουθήσουμε, την ε, ε, κοινή γεωργική πολιτική σε συνδυασμό και με την αλλαγή του κλίματος και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και επίσης θα πρέπει να απαντήσουμε στις ευρύτερε ανησυχίες ε, για το ευρύ κοινό. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε υψηλής ποιότητας τρόφιμα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Προσβλέπω στην ε, συνεργασία με την Προεδρία σας για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις συζητήσεις. Εμείς τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να προωθήσουμε τις συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή μας και να παρουσιάσουμε ε, μία εικόνα που αντιπροσωπεύει την άποψη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τι μελιγενέστε. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Ο, ο κύριος Χάουσλινγκ. Ναι, Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Ε, ουσιαστικά λέτε ότι στο Συμβούλιο η... ο διχασμός και οι διαφορετικές απόψεις είναι εξίσου διαφορετικές όπως και στο Κοινοβούλιο και ότι υπάρχει ανάγκη να συζητήσουμε πρωτού καταλήξουμε στη συνένεση και σε τελική ανάλυση ελπίζουμε να εφαρμοστούν τα όσα αποφασιστούν στο, για την αγροτική πολιτική. Να υπάρχει και η τόλμη από πλευρά Συμβουλίου να εφαρμοστούν όλα όσα θα αποφασιστούν. Υπάρχουν κάποια αμφιλεγόμενα σημεία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο το θέμα των ανώτατων ορίων, για παράδειγμα, αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί αποτελεί και ένα ζήτημα ε, ισότητας της κατανομής και θα πρέπει να ασχοληθούμε επίσης με το τι σημαίνει ότι οι γεωργοί συμμετέχουν στην διατροφική αλυσίδα με, υψηλή, με υψηλό κέρδος. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα και ελπίζουμε να ακολουθήσουν σωστές προτάσεις από το Συμβούλιο. Χάρηκα και που αναφέρατε το θέμα του πρασινίσματος. Ε, θεωρώ ότι αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, δεν αποτελεί τα δευτερεύοντα στοιχεία της αγροτικής πολιτικής. Θα αποτελέσει θέμα κλειδί. Και θα πρέπει έτσι να δικαιολογηθούν και οι δαπάνες για την αγροτική πολιτική. Να σας πω ότι χτες παρουσιάστηκε μία μελέτη ότι υψηλή, το υψηλό ποσοστό αζότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλείται κυρίως από τη γεωργία και αυτό συνεπάγεται τεράστιο κόστος. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με κριτικό πνεύμα σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της εντατικής καλλιέργειας. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο στην Ευρώπη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα περιβαλλοντικά μέτρα και ελπίζω να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση στο Συμβούλιο στην περαιτέρω συζήτηση. Ο κύριο και μετά ο Στεφάν Λεφόλ. Η κυρία συγγνώμη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον Υπουργό Φαζέκα και θα ήθελα να ρωτήσω σε εκπρόσωπος της Προεδρίας και υπό την ιδιότητά του ως υπουργός της χώρας μου. Ε, θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να διευκρινίσω κάποια ερωτήματα βασικά σχετικά με τις ε, θεμελιώδεις αξίες και είναι αυτό το πνεύμα που υπέβαλα τις τροπολογίες μου στην έκθεση. Πρώτη ερώτηση κάπως τεχνική. Προτείνω μία ονομασία, κοινή πολιτική ονομασία της ε, γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιο πως αμυδρή διαφορά, αλλά είναι θέμα ουσίας. Θέλουμε να διατηρήσουμε την το αγροτικό περιβάλλον. Δεύτερο ερώτημα που σχετίζεται με το πρώτο, και έχει να κάνει με την φύση του συστήματος ενισχύσεων που θα θεσπίσουμε. Θα εξαρτάται από αυτό το σύστημα, θα, θα, θα εξαρτάται από το εάν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν στις αγροτικές περιοχές. Μήπως ο υπουργό είναι υπέρ της εισαγωγής ενός πλαφών, ενός ανώτατου ορίου για τις εκταρικές πληρωμές. Νομίζω είναι άδικο οι φορολογούμενοι, οι Ούγγροι και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να χρηματοδοτούν τον πλουτισμό των ε, δισεκατομμυριούχων που που ζουν από την γεωργία και που χρησιμοποιούν πολύ χαμηλά εργατικά. Για τους ε, Ούγγρους ε, ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν άτομα που ε, παίρνουν 300 εκατομμύρια ε, ενισχύσεις αγροτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας ε, τραπεζίτης στη Βουδαπέστη που δεν ξυπνάει πολύ νωρί το πρωί να δουλέψει τη γη. Είστε υπέρ της εισαγωγής ενός ανώτατου ορίου και η Ουγγρική Προεδρία και εσείς Υπουργέ είστε υπέρ της εισαγωγής μίας ε, ελάχιστης ε, πληρωμής που να επιτρέψει στους αγρότες, τους μικρούς και νέους αγρότες να επιβιώσουν στις αγροτικές περιοχές ή σε νέους να μπουν στον αγροτικό τομέα. Τρίτη ερώτηση, ποια είναι η άποψή σας ε, κύριε Υπουργέ για το θέμα, το σφαιρικό θέμα του το, παγκόσμιου εναντί τοπικού Πιστεύετε ότι τα καλά προϊόντα είναι αυτά που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Ε, θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η λειτουργία των μικρών μεταποιητών, μικρών παραγωγών ε, τροφίμων και αγροτικών ε, προϊόντων. Τελευταία ερώτηση, πιο συγκεκριμένη τώρα, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε και σε αυτό το θέμα. Συμφωνείτε κύριε Υπουργέ ε, για την απαγόρευση απλά και μόνο των εισαγωγών προϊόντων που δεν ε, συνάδουν με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών που είναι αυστηροί. Ούγγροι γεωργοί θα πρέπει να τηρούν αυτούς τους αυστηρούς κανόνες, αλλά η πλειοψηφία των παραγωγών του τρίτου κόσμου δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες. Είναι άδικο. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη είναι σημαντική αξία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επισέλθω στη συζήτηση Ουγγρών, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν θα δω κατά πόσο εσείς ξυπνάτε πρωί για να ε, δουλέψετε τη γη, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα μόνο. Θα πρέπει να έφτασε τώρα η μετάφραση στα Ουγγρικά, φαντάζομαι. Ε, την παρουσίαση για τη δουλειά του Συμβουλίου, για τους στόχους, συμφωνούμε θα πρέπει να έχουμε στόχους ε, μιας πολιτικής, μιας αγροτικής πολιτικής που είναι ανταγωνιστική βέβαια, βιώσιμη και που να λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό, την κοινωνική πτυχή της γεωργίας σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. Θα πρέπει αυτή η γεωργία και η ΚΑΠ είναι το λέμε ισότιμη δίκαιη στην κατανομή των πόρων και θα πρέπει να είναι η φόρο. Στο θέμα αυτό, ο Άλμπερτ που έχει δουλέψει πολύ σκληρά, όπω το ξέρουμε εμεί εδώ στην Επιτροπή μα, πρότεινε συμβιβασμού. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο τη παρουσίαση που θα κάνει αργότερα. Αλλά είμαστε υπέρ, ε, όπως το Κοινοβούλιο, να ε, ε, ορίσει μια θέση κατόπιν τη της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, έχετε χαιρετήσει αυτή την ανακοίνωση και εμείς πάμε προς την κατεύθυνση αυτής της ανακοίνωσης και θα ήθελα να ρωτήσω μια ερώτηση σε αυτό. Στο Συμβούλιο συζητήσατε το θέμα της αηφορίας της γεωργίας ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα. Έγινε κάποια συζήτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια πρόταση που να μην είναι αυτή που παρουσιάστηκε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο στην ανακοίνωσή του. Μήπως αναφέρθηκε για παράδειγμα ότι θα έπρεπε να τροποποιήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα για θέματα περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ Στεφάνο. Κύριος Νίκολσον. Κυρία Μορβέη, Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσατε να πείτε στον εκπρόσωπο της Τράπεζας των Εκατομμυριούχων, γιατί φαντάζομαι ότι αυτούς εκπροσωπείτε, να το ξέρουν οι ψηφοφόροι σας ότι τους εκπροσωπείτε, ότι εκπροσωπείτε εκατομμυριούχους τραπεζίτες, Καταρχάς να βελτιώσετε λίγο την αίσθηση του χιούμορ σας και να διατηρήσετε τις προσωπικές σας παρατηρήσεις για τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ας το ευχηθούμε όλοι, λέει ο Πρόεδρος. James, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Υπουργό, εδώ σήμερα το απόγευμα. Γνωρίζετε ότι είχαμε τη δυνατότητα να μεταβούμε στην Ουγγαρία πριν από τα Χριστούγεννα και επειδή πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην Ουγγαρία τα είδαμε η σώμαση. Ήταν σημαντικό άλλωστε αυτό, διότι κάποιοι από τα παλιά κράτη-μέλη μπόρεσαν να διαπιστώσουν πόσο διαφορετικά είναι τα προβλήματα των νέων χωρών μελών. Νομίζω ότι το βασικό που θα έχουμε για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το θέμα του πρασινίσματος της γεωργίας. Εγώ έχω πολύ στεναρή άποψη. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πρασίνισμα στον πυλώνα 1 σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι οι αρμοδιότητε του πυλώνα 2 είναι μια χαρά για να υποστηρίξουμε τα θέματα και το ξέρω ότι περισσότεροι υποστηρίζουν διαφορετική άποψη και τη σέβομαι. Πιστεύω ότι το συζητάμε πολύ και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Όλο λέμε ότι θα πατάξουμε τη γραφειοκρατία, ότι θα σταματήσει το γραφειοκρατικό άκθο και θα είναι η διασταυρούμενη συμμόρφωση πιο εύκολη για του γεωργού για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του. Και παρά το γεγονό ότι όλοι μιλάνε για πράσινου όρου, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι όποια απόφαση και αν λάβουμε, όποια οδηγία και αν περάσει, σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, περισσότερη γραφειοκρατία. Πώς θα το καταλήξουμε αυτό, πότε θα το σταματήσουμε, πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα τέλος για όλους. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι στη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και στην έκθεση DES. και ο Επίτροπος, βέβαια δεν έχω και μεγάλες προσδοκίες, αλλά ελπίζω ο Επίτροπος όταν παρουσιάσει το νομικό του κείμενο στο τέλος ε, του έτους να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Να σας πω επίσης ότι ακούσατε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εν τέλει όλοι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία θέση. Κανένας μας δεν θα τα πάρει όλα ως επιθυμεί, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει και θα έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που θα είναι αποτελεσματική και θα μας δώσει αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μας. Και θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια θέματα. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για τους επόμενους μήνες προς το τέλος ε, της Προεδρίας σας για τα γαλακτοκομικά, αλλά ε, θεωρώ ότι κάποια από τα πράγματα θα έπρεπε να προκύψουν ήδη από τώρα. Ε, δεν μπορούμε να ε, κολλήσουμε στον τοίχο τους μικρούς γεωργιούς και να τους αποτρέψουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, όπως και αν το αντιμετωπίσουμε, θα υφίσταται πάντα και πρέπει να βρούμε μία λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, James, ο κύριος Άγνιου και μετά ο κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τεχνική ε, ερώτηση που θέλω να θέσω προς τον ε, ε, Υπουργό. Μας είπατε σύγκληση. Αυτός, ξέρετε, είναι λίγο φορτισμένο όρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί θεωρούμε ότι η σύγκληση σε αυτό το επίπεδο αποτελεί την εξίσωση των πληρωμών για τα κράτη-μέλη, τα παλιά και τα καινούργια. Και από ό,τι ξέρετε, τα παλιά κράτη-μέλη στην παρούσα φάση παίρνουν πιο πολλά. Η σύγκληση λοιπόν τι σημαίνει για πολλούς από εμάς, εξίσωση, ισοπαίδωση. Ξέρω ότι μερικοί μερικοί μόνο το ε, καλωσορίζουν αυτό, αλλά πολλοί από τους ε, Βρετανούς φορολογούμενους θα χάσουν. Το άλλο που μπορεί να σημαίνει η σύγκληση είναι η σύγκληση των απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο μπορεί να εννοούσατε, θα μπορούσατε όμως να το διευκρινίσετε. Ίσως θα μπορούσατε να μιλήσετε και για την εξίσωση αυτή των πληρωμών. Ευχαριστώ. Ντόρφμαν και μετά Γκαρσία Περέση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ σήμερα για να μας παρουσιάσετε τη θέση του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής. Νομίζω ότι τα πιο πολλά από αυτά που είπατε μας βρίσκουν σύμφωνους. Γρήγορα να διατρέξω κάποια σημεία. Μιλήσατε για την κατανομή, την ανακατονομή των άμεσων πληρωμών, όπου σας δίνω απόλυτο δίκιο θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό δεν ισχύει όμω μόνο σε ό,τι αφορά την κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά την κατανομή στο εσωτερικό των κρατών μελών. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι από ένα κράτος μέλο από την Ιταλία, όπου μεταξύ των περιφερειών της ε, χώρας υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν πιο πολλές άμεσες πληρωμές και υπάρχουν και άλλες που λαμβάνουν πολύ λιγότερες. Αυτό έχει να κάνει με τις ιστορικές, ε, με τους ιστορικούς υπολογισμούς. Νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός να αφήσουμε τους ιστορικούς ε, υπολογισμούς και να κοιτάξουμε την επιφάνεια. Μιλήσατε για να τα όρια επίσης. Νομίζω ότι οι πληρωμές στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να αποτελούν και μία αποζημίωση σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ανώτατα όρια, θα πρέπει να υπάρξει μία λύση, γιατί δεν υπάρχει αφιβολία ότι η επεξεργασία ε, μεγάλων επιφανείων είναι, εκτάσεων είναι πιο ακριβή για μικρές επιχειρήσεις από ότι για μεγάλες. Αυτό αποτυπώνει την κατάσταση και το κόστος της γεωργίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να ακολουθήσουμε άλλες λύσεις πέρα από την ε, ανώτατη από τα ανώτατα όρια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά τεχνική λόγη για την ε, εφαρμογή ανώτατων ορίων. Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσυμφορηθούν σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθος και πιο πολύ θα τις βοηθούσαμε αν απλοποιήσουμε το σύστημα αποτελεσματικά, παρά με πολλά άλλα μέσα τα οποία προτείνονται εδώ. Κλείνοντας, να πω και δύο λόγια για το γάλα το οποίο αναφέρατε. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφώς σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται, αλλά δεν δίνει απάντηση για την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015. Ιδιαίτερα στις δύσκολες ορεινές περιοχές, η κατάργηση των ποσοστώσεων για το γάλα θα σημαίνει σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν σε επίπεδο αγροτικής πολιτικής να σκεφτούμε πώς μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή τέτοιες γαλακτοκομικές επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές. Γιατί αν καταργηθεί ουσιαστικά η γαλακτοπαραγωγή καταργείται το σύνολο της γεωργίας σε τέτοιες ε, περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό, προκειμένου πριν καταργηθούν οι ποσοστώσεις να δούμε τι θα γίνει, προκειμένου να υπάρχει ένα μέλλον για τις επιχειρήσεις αυτές. Ευχαριστώ, κυρία Γκαρσία Πέρες. Μετά ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, κάνω μια σύνδεμη αναφορά στην έκθεση του κυρίου Ντες ε, για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο πακέτο στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος. Γνωρίζετε ότι εχθές έγινε η παρουσίαση της έκθεσης και η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλά προβλήματα θα μπορέσουμε να έχουμε κοινή θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν το Συμβούλιο να δείξει διάθεση για συνεργασία προκειμένου να λάβει υπόψη και τις ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα όσα θέλουμε να έχουμε στο πακέτο ποιότητας, ε, κυρίως όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, τον καλύτερο ορισμό ε, αυτών και ούτω καθεξής. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παρούσα συνεργασία και να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ε, παρόν σύστημα προστασίας της ποιότητας. Όσον αφορά τώρα την έκθεση του κυρίου Ντές, ε, τόσο ο συντονιστής ο κύριος Καπούλας ε, Σάντων, όπως επίσης και ο σκιώδης εισηγητής των σοσιαλιστών, ο κύριος Λεφόλ, παρουσίασαν τις θέσεις της ομάδος για την έκθεση αυτή. Είναι αλήθεια ότι έγινε μια προσπάθεια με στόχο να έχουμε μια κοινή θέση και να προασπίσουμε κοινέ αρχέ. Όπω και ο, ο του Συμβουλίου, όπω και εμεί θεωρώ ότι συμφωνούμε για τι βασικέ γενικέ αρχέ, ούτω ή άλλως τις συζητάμε εδώ και ένα χρόνο, τι προκλήσει, ε, τι ε, λήψει και ούτω καθεξή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική, θέλουμε οικονομική ενέσχυση, είναι πολύ σημαντικοί οι δύο πυλώνες, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία θα πρέπει η Επιτροπή μας αλλά και οι υπεύθυνοι των πολιτικών ομάδων να κάνουν μια προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κοινό σημείο και να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα συμβιβασμό στον οποίο θα καθορίσουμε όλοι τους στόχους μας. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτόν ακριβώ το λόγο να αναφερθώ σε δύο θέματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Καταρχά υπάρχει το θέμα των νέων, νομίζω ότι αποτελούν σημαντικό και θεμελιώδη παράγοντα, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίση ότι και οι γυναίκε είναι σημαντικό παράγοντα για την ε, ανάπτυξη τη υπαίθρου και θα πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία ενίσχυση στην κοινή γεωργική πολιτική για να έχουμε και ένταξη των γενικών και συμμετοχή τους ε, και στις γεωργικές ε, ε, εκμεταλλεύσεις και στις γεωργικές εργασίες αλλά και στην ανάπτυξη της υπαίθρους. Όσον αφορά τώρα τους νέους και τις άμεσες, ε, ισχύει το ίδιο. Τώρα για τις άμεσες ε, επιδοτήσεις, τις άμεσες ενισχύσεις, νομίζω ότι κανείς εδώ στην Επιτροπή δεν μπορεί να είναι κατά της βασικής αρχής, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όταν ε, θα ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του μέσου των άμεσων ενισχύσεων και θα πρέπει να λάβουμε υπέψη και τις μεταβατικές περίοδου, περιόδους. Τις έχουμε πολλοί από εμάς τοποθετήσει στον πρώτο πυλώνα. Επίσης, όταν αναφερόμαστε στην ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας, ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και όταν μιλάμε για τις μεθόδους κτηνοτροφικής παραγωγής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μεθόδους κτηνοτροφικής παραγωγής χωρίς ε, ε, γεωργικές εκθάσεις. Πρόκειται για μια μορφή παραγωγής που, δεν, που είναι πολύ διαδεδομένη στη Μεσόγειο και υπάρχουν πολλά προβλήματα στο συγκεκριμένο τομέα, στο κτηνοτροφικό ε, αντιμετωπίζονται προβλήματα και χρειάζεται μεγαλύτερη όθηση μέσα στήριξη και να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές και να λάβουμε υπόψη και την κτηνοτροφία αυτή χωρίς ε, χερσαίες εκτάσεις. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ κύριος Γιάρ και μετά ο Ζωζεμποβέ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τόνισαν όλοι οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες, ότι υπάρχουν ε, και συμφωνίες, ε, ευρεία συμφωνία μάλιστα. Όλοι είμαστε υπέρ της αγροτικής ε, πολιτικής, θέλουμε σωστή χρηματοδότηση, είμαστε υπέρμαχοι της στρατηγικής των δύο πυλώνων, θέλουμε ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, βιωσιμότητα. Συμφωνούμε ευρέως για το πρασίνισμα, όπως ονομάζεται, της γεωργίας. Και διαφωνούμε, μάλλον ε, συμφωνούμε και για την ε, απλούστευση. Να ευχαριστήσω και την προηγούμενη ομιλήτρια γιατί μίλησε για την ε, διαφοροποίηση. Εγώ είμαι από τη Γερμανία, όπου έχουν αναπτυχθεί οι δομές που έχουν αναπτυχθεί, όχι εντελώ εθελούσια, αν το λάβουμε υπόψη αυτό. Οι γεωργοί μας ε, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση το 60 και το 90 αποφάσισαν ε, ότι θα ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή και αποφάσισε μεγάλο τμήμα των γεωργών να συνεχίσει μαζί την παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι κάπως πιο μεγάλες από τις άλλα τμήματα της Ευρώπης, γιατί ε, ε, έγιναν ενώσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις τρέφουν και πολλές οικογένειες. Και όταν ε, στην περιοχή μου είχε έρθει η σοσιαλιστική, ο σοσιαλισμός και είχε επιβάλει κάποια στοιχεία. Τώρα επιβάλλει η πολιτική κάποια άλλα στοιχεία, κάποια διαφορετική πολιτική. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι της, Ευρω... της γεωργικής πολιτικής. Περιβαλλοντική προστασία, ανταγωνιστικότητα. Αν αυτή είναι η στόχη μας, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναπτύξουμε και ε, συγκεκριμένες δομές οι οποίες να γίνουν αποδεκτές. Σας παρακαλώ λοιπόν όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα και συζητάμε μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις Κοιτάξτε σε εμά σε γενικέ γραμμέ ο διευθυντή μια ε, αγροτική ένωση και αυτός πρωί σηκώνεται. Να μην του καταστρέψουμε λοιπόν. Τελευταία παρατηρήση. Δεν έχει νόημα η πολιτική να προδιαγράφει και το μέγεθος της επιχείρησης γιατί σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε και την ανάλογη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο Ζωζέ Μποβέ και μετά ο κ. Ρένα. Θα ήθελα να παρέμβω σε τρία σημεία. Ξεκινώντας από μια πραγματικότητα και έχουμε ήδη ακούσει και προηγουμένως κάτι σχετικό. Στην Ευρώπη οι λαϊκισμοί και τα κίνηματα τα ξενοφοβικά δυστυχώς αυξάνονται με ένα κίνδυνο για την δημοκρατία φυσικά. Και αυτά τα κινήματα συχνά αναπτύσσοντας ε, με βάση τις αδικίες που υπάρχουν και επιδεινώνοντας αυτή την κατάσταση στην συζήτηση. Είδαμε πως ε, μια ε, αντιπρόσωπο ενός μια ξενόφοβου ομάδας. Αν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή την κατάσταση και δεν κάνω οποιαδήποτε επίθεση σε άτομα. Όλα, όλοι οι βουλευτές είναι ήδη σε αυτή την συνέλευση. Αλλά πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις συμπεριφορές. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η αδικία, η, δικαιοσύνη, με συγχωρείτε. Και αυτή είναι σημαντική στην ΚΑΠ. Είναι η μόνη ολοκληρωμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θέλουμε αυτή η δικαιοσύνη να υπάρχει και αν θέλουμε να αποφύγουμε εθνικιστικές κινήσεις, θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στα κράτη και να, να κατανέμεται ισότιμα να κατανοούνται ισότιμα οι ενισχύσεις ανάμεσα στα κράτη, ανάμεσα στις περιφέρειες. Θα πρέπει να υπάρχει η δικαιοσύνη είναι ανάμεσα στι περιφέρειε, διότι υπάρχουν ευνοούμενε και λιγότερο ευνοούμενε ε, περιφέρειες. Δικαιοσύνη ανάμεσα στου γεωργού. Αυτό είναι σημαντικό στην κατανομή των ενισχύσεων, διότι δεν μπορεί το 75% των ενισχύσεων να κατανέμεται σε 25% των γεωργών. Αυτή είναι η βάση της μεταρρύθμισης και εδώ αναφέρομαι και στον κύριο Ντες, διότι πρέπει αυτό το κοινοβούλιο να έχει μια κοινή θέση για να επιβεβαιώσουμε αυτό το κοινό βάρο η Ευρώπη χωρίς τη γεωργία δεν υπάρχει. Η Ευρώπη η γεωργική είναι η Ευρώπη όλων των γεωργών αλλά και των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. Ο κύριος Ρέμε, Ευχαριστώ και χάρηκα που ήρθατε σήμερα στη συζήτηση. Ο κατάλογος που μας δώσατε σε ό,τι αφορά τις θέσεις του Συμβουλίου με απασχολεί κάπως. Γιατί είναι εξίσου μακρύς όπως και ο δικός μας κατάλογος. Έχουμε όλοι πολλές επιθυμίες για την αγροτική πολιτική. Κανείς όμως δεν έχει λύσεις για να τη χρηματοδοτήσει τη λύση αυτή. Νομίζω ότι η μεγάλη συζήτηση είναι πως όλες αυτές οι λύσεις θα χρηματοδοτηθούν με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω λοιπόν ότι ο καιρός είναι να κάτσουμε και να συζητήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Τι είναι το πιο σημαντικό το οποίο θα πρέπει η πάση θυσία να χρηματοδοτηθεί και πού μπορούμε να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι ίσονος σημασίας. Όλοι ξέρουμε, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ότι κανείς δεν θέλει να πληρώσει παραπάνω. Όμως όλοι θέλουμε πιο πολλά καθήκοντα, πιο πολλούς στόχους. Αυτό μαθηματικώς πώς δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ειλικρινεί έναντι και των γεωργών και να πούμε ότι κοιτάξτε αυτό είναι η προτεραιότητά μας και όχι το χύψη. Παρά να παρουσιάζουμε όλοι οι καταλόγους με σκοπό να ικανοποιήσουμε τους πάντες, αλλά χωρίς να είμαστε ρεαλιστές. Ευχαριστώ λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας ε, μιλήσατε για τις εργασίες του Συμβουλίου. Θα ξεκινούσα με το τελευταίο θέμα το οποίο γύρατε, το πακέτο γάλα και ποιότητα. Μας κάνετε μια πρόταση συνεργασίας ε, για να κλείσουμε σε πρώτη ανάγνωση υπό Ουγγρικής Προεδρία. Νομίζω είμαστε σύμφωνοι με αυτό. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να συζητήσει δύο ή τρία θέματα που είναι κάπως διαφορετικά. Έχουμε εκφραστεί ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης της ε, παραγωγής για τις ονομασίες ε, ε, στις ορεινές περιοχές. Ελπίζω να υπάρχει καλή συνεργασία. Στην ΚΑΠ μας δώσετε ένα μακρύ κατάλογο των θεμάτων που θέλει να λάβουμε υπόψη στο Συμβούλιο, αλλά δεν μας μιλήσατε για χρήματα. Και ο πρόεδρος Βαρόσο θα πρέπει να παρουσιάσει υπό Ουγγρικής Προεδρίας το σχήμα του προπολογισμού για την μελλοντική περίοδο. Μπορείτε να μας δώσετε την άποψη του Συμβουλίου στο θέμα αυτό, το δημοσιονομικό, του προϋπολογισμού. Ε, το Κοινοβούλιο εκφράστηκε ε, επιθυμώντα τη διατήρηση του προπολογισμού στο επίπεδο που υπάρχει. Το ίδιο αναφέρει και ο Αλμπερντές, τι άποψη έχει το Συμβούλιο και επειδή εκπροσωπείται και την Προεδρία, ποια είναι η άποψη της Ουγγρικής Προεδρίας για τι δημοσιονομικέ προοπτικές και κυρίω για τη θέση τη γεωργία της δημοσιονομική προοπτική τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε Μισελ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχετε εσείς το λόγο και έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στις διάφορες παρεμβάσεις. Θα ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ και ελπίζω να μπορέσετε να εργαστείτε όπως αποδείξαμε σήμερα το απόγευμα σε κλίμα συνεργασίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μα απευθύνατε τις ερωτήσεις σας. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία συνεργασίας και είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον της ΚΑΠ προς το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών για να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι εμφανές ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πολλές διστάμενες και διαφορετικές απόψεις, διότι η Ευρώπη είναι μια ε, ε, περιφέρεια και μια περιοχή της ποικιλομορφίας. Το ίδιο και η γεωργία. Το πιο σημαντικό είναι να ε, προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και αυτή η κατεύθυνση πρέπει να είναι η κατεύθυνση της ισχυρής Ευρώπης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και αν ε, είναι μακρύς ο κατάλογος των ερωτήσεων. Προς τον κύριο Ντές ξεκινώ τον κύριο Κάπουλας Σάντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προτάσεις συνεργασίας τους και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τις απόψεις τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που θα επιτρέψουν να ε, έχουμε μία παραγωγική και αηφόρο γεωργία και θα βρούμε ένα σύστημα ενισχύσεων. Ε, φυσικά η ΚΑΠ δεν είναι απλά μία μάζα νομοθετικών πράξεων. Η ΚΑΠ έχει αποδείξει την νομιμότητα της εδώ και πολλά χρόνια και χρειαζόμαστε πάντα ε, την ΚΑΠ για να διασφαλίσουμε μια επισητιστική ασφάλεια μακροχρόνια. Τώρα, στο θέμα του πρασινίσματος ε, προς τον κύριο Λάιονς και σε άλλους που θέσανε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα που ανησυχούν ε, ε, βέβαια και την κοινή γνώμη. Το σημείο 16 των συμπερασμάτων τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απλή λύση και όχι δαπανηρή για να διασφαλιστεί ο στόχος η περιβαλλοντική στόχη μάλλον. Θα πρέπει το σύστημα ενισχύσεων να στηρίζεται σε περιβαλλοντικές πτυχές και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να σκεφτούμε τις ε, κλιματικές αλλαγές, τη διαχείριση των υδάτων. Δηλαδή δεν θα σταματήσουμε στο ε, πώς θα είναι η ε, κατανομή ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Ήδη στο πρώτο πυλώνα υπάρχουν στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον και βεβαίως στο δεύτερο πυλώνα θα ενισχυθούν αυτά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποκλήσεις στις απόψεις των κρατών μελών στα θέματα αυτά. Τώρα, στο θέμα της ε, παραγωγής ε, τροφίμων καλής ποιότητας μπορεί να αποκαλέσουν κοινωνικά προβλήματα. Δεν κατάλαβα πολύ καλά το νόημα της ερώτησης. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη έχει την ε, ε, παραγωγή τροφίμων βέλτιστης ποιότητας, της καλύτερης στον κόσμο και αυτή η παραγωγή καλής ποιότητας διασφαλίζεται και από το σύστημα ονομασίας προέλευσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε ένα επίπεδο απασχόλησης ε, τον τομέα τον γεωργικό. Στα συμπεράσματα επίσης τονίσαμε την σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου, της αγροτικής ανάπτυξης. Προς την κυρία Μορβάη, θα ήθελα να απαντήσω ότι η ονομασία μπορεί να αλλάξει μελλοντικά. Έχουμε ξεκινήσει από το σημείο ότι η ΚΑΠ ονομαζόταν Κοινή Αγροτική Πολιτική. Άρα με αυτό εννοούμε κάτι ευρύτερο από το περιορισμένη, την περιορισμένη έννοια του όρου. Ε, εννοούμε επίσης μια περιβαλλοντική πολιτική, μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Στο θέμα της, ε, των ορίων, ανωτά των ορίων των ενισχύσεων έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα ε, στο θέμα αυτό. Βέβαια υπάρχει αντίσταση εκ μέρους των κρατών μέλων για να τεθούν ανώτατα όρια στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε ακούσει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και χωρίς να διακυβεύεται η απλούστευση της ΚΑΠ. Πιστεύω ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά της θέσης ανωτά των όριων και ε, υπάρχουν δίσταμνες απόψεις. Ε, νομίζω ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις στον τομέα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο στα κράτη-μέλη, διότι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν μικρές εκμεταλλεύσεις και αυτό που θα ήταν επιθυμητό ήταν αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις να γίνουν μεγαλύτερες, μεσαίου μεγέθους και μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Βέβαια αυτό το ερώτημα συνδέεται και με το θέμα των νέων γεωργών, των νέων αγροτών. Και είναι επίσης ε, σίγουρο ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, λύσεις που να υποφελούν ε, διάφορα αρκετά Τώρα, το θέμα της ποιότητας, καλής ποιότητας τροφίμων και τοπικής παραγωγής, αυτό υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη και από την Ουγγρική Προεδρία από ε, την άποψη των καταναλωτών και του περιβάλλοντος είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Ταυτόχρονα επιτρέπει τη διασφάλιση των παραδοσιακών προϊόντων. Στο πακέτο ποιότητα ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Στο θέμα των εισαγωγών από τρίτες χώρες υπάρχουν βέβαια διεθνείς συμφωνίες και δεν μπορούμε απλά να τις παραβλέψουμε. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Θα ήθελα απλά να υπογραμμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα και των γεωργών και των Ευρωπαίων καταναλωτών πάνω απ' όλα. Τώρα, στο θέμα του, που έθεσε ο κύριος Λεφόλ, συμφωνώ απόλυτα ότι η αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι δίκαιη και δίκαιη αλλιώς δεν έχει μέλλον. Σε ό,τι αφορά την κατανομή ανάμεσα στους δύο πυλώνες, αυτό συνδέεται με το θέμα της αηφορίας και του τομέα στον οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε την, την γεωργική παραγωγή. Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Το έχει συζητήσει ήδη αυτό το θέμα. Επήρξαν και άλλα ερωτήματα σχετικά με το πρασίνισμα. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα θα πρέπει να μειώσουμε το χαρτοβασίλειο, τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο παρελθόν. Κάθε φορά που θέλαμε να απλουστέψουμε το σύστημα, τελικά το περιπλέκαμε περισσότερο. Θα πρέπει να εναρμονιστούν οι απόψεις. 26 κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει μια ανακοίνωση, ένα ανακοινωθέν σχετικά με τις, τους προσανατολισμούς της διοικητικής απλούστευσης. Τώρα, στο θέμα που έχει σχέση με την σύγκληση, το σημείο 9 των συμπερασμάτων περιλαμβάνει τα εξής. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να κατανέμονται με πιο ισορροπημένο τρόπο ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να μειώσουμε σταδιακά την σύνδεσή τους με την προηγούμενη αναφορά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης το γενικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο έχετε εξασφαλίσει την απάντησή σας. Το Συμβούλιο κατόρθωσε να ε, πετύχει ένα συμβιβασμό σε αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια είναι πολύ περίπλοκο θέμα, διότι οι συνθήκες ε, οι δημοσιονομικές, των τιμών, τις παραγωγές, όλες αυτές διαφέρουν ακόμη και σε, στο κάθε κράτος μέλος μέσα. Όταν μιλάμε για ισότιμη κατανομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να δοθεί χώρος κίνησης και ελιγμών σε κάθε κράτο μέλος για να εξασφαλίσουν αυτή την ανταγωνιστικότητα. Στο θέμα των μικρών γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων. Ο κύριος Ντόρφμαν αναφέρθηκε στις ορεινές περιοχές. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι σε αυτές τις περιοχές δεν ε, θα μπορούσε να υπάρχει απασχόληση χωρίς τον καλαχτοκομικό τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το θέμα στο πακέτο γάλα που είναι θέμα προτεραιοτήτων υπό Ουγγρικής Προεδρίας. Στο θέμα που έφτιαξε η κυρία Γκαρσία Πέρες σχετικά με το πακέτο ποιότητας, είμαι αισιόδοξο ε, σε αυτό το μέτωπο. Ε, πιστεύω ότι αυτό που είπατε ενισχύει το δικό μας προσανατολισμό. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύοντας την προστασία των καταναλωτών και ενισχύοντας επίσης την αγροτική πολιτική. Έχουμε ήδη αποτελέσματα τα οποία το καταδεικνύουν. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των νεαρών ε, αγροτών, ε, είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση του Κοινοβουλίου χωρίς νέους, χωρίς γυναίκες, δεν μπορεί να υπάρξει γεωργία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το ζήτημα. Τώρα, για να απαντήσω στην κυρία Ρέμερς. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση, είναι κρίσιμη σημασία το ερώτημα. Μιλάμε για γεωργική πολιτική η οποία απαιτεί εργαλεία, μέσα. Εμείς ορίζουμε τους στόχους, τους έχουμε ήδη ορίσει στα συμπεράσματα της Προεδρίας. Πρέπει αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν μέσα από την αγροτική πολιτική και στο επόμενο στάδιο θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για το χρηματοδοτικό πακέτο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά αυτό την προσοχή σας στο σημείο 4 των συμπερασμάτων που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό μια ισχυρή ΚΑΠ, η οποία θα έχει τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είναι αναλογικά ως προς τους στόχους. Πράγμα που καταδείκνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Για να απαντήσω στον κύριο Νταντάν που έθεσε το ερώτημα σχετικά με το πακέτο του γάλακτος και της ποιότητας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τον γαλακτοκομικό τομέα, διότι είναι ένας τομέας ε, εμβληματικός, σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό του δίνουμε προτεραιότητα στη διάρκεια της δικής μας προεδρίας, στον τομέα του γάλακτος. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Προσπάθησα να απαντήσω με συντομία. Ε, είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και ότι θα πετύχουμε και θα καταλήξουμε σε όλα αυτά τα δοσιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φαζέκας ε, και για τη διαθέσιμά του και για την ενημέρωσή του. Ένα λεπτό διακοπή για να χαιρετήσουμε τον ε, Υπουργό και να συνεχίσουμε στη συνέχεια με το σημείο 13. Prendiamo posto. Καθίστε παρακαλώ. Prendiamo posto. Καθίστε παρακαλώ. is there. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Καλώς. Να περάσουμε τώρα στη συζήτηση για το σημείο 12. Άλμπερτ, να ξεκινήσουμε Λαμβάνοντα υπόψη ότι σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα Δεδομένου ότι έχουμε και 1.267 τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν στο σχέδιο έκθεσης του Αλμπερντές για την κοινή αγροτική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν και οι συντονιστές αποφάσισαν να αναβληθεί η ψηφοφορία της ε, έκθεσης αυτής για τις 25 Μαΐου, αντί για τις 2 Μαΐου. Βέβαια, στο μεταξύ έχουμε πολύ σημαντική δουλειά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Άλμπερτ μαζί με όλους τους κοιόδης εισηγητές θα εργατιστούν εντατικά αυτές τις μέρες προκειμένου να μπορέσουν να συμπυκνώσουν σε λίγες συμβιβαστικές τροπολογίες ε, τα θέματα αυτά όπως κάναμε και με την ε, προηγούμενη έκθεση Lion. Τώρα, επειδή είναι πολύ σημαντικό το εργαστήριο που έχουμε μετά από αυτή τη συζήτηση, αν συμφωνείτε θα ήθελα μετά από την παρέμβαση του Albert να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι ο Διευθυντής, ο Τάσος Νιώτης, ε, θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ ή αν δεν είναι, είναι καθοδόν και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης εισηγητές για να γίνει μια πολύ... Ε, μια συζήτηση συγγνώμη, που θα είναι επικεντρωμένη κυρίως ε, στην έκθεση, να μην καθυστερήσουμε πολύ και να υπάρχει και περιθώριο για πιο εις βάθος συζήτηση. Έχουμε εδώ τους ε, ε, εμπειρογνώμονες, ε, τον David Baldock και τον και Albert Wildman και τον Κοράντο Λιτιτσέτο και αν είστε έτοιμος Albert, ο κύριος Παπαστάμκος έχει ζητήσει το λόγο. Είτε, αλλά γιατί δεν προτάσσονται τα σύντομα τα θέματα το υπαρίδουν 15 και 16 να τελειώνουμε αυτά για να έχουμε όλο το χρόνο για την ε, έκθεση του κυρίου Ντές που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Διαφορετικά φοβούμε ότι δεν θα μείνει καθόλου χρόνος και ενώ αυτό θα είναι πέντε λεπτά οι συζητήσεις. If. Okay. Ε, έχεις δίκιο Γιώργο. Μάλλον δεν θα μας μείνει πολύ ώρα για να τα συζητήσουμε αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θα πρέπει να φύγουν, εγώ θα ήθελα να προτείνω στη γραμματεία να τις αναβάλουμε τις συζητήσεις για τα 15 και 16. Είναι πολύ γρήγορα τα θέματα. Αν δεν τα κάνουμε σήμερα, μπορούμε να το κάνουμε και στην επόμενη συνεδρίαση και να αφιερώσουμε το χρόνο που έχουμε σήμερα το απόγευμα στα δύο σημεία 12 και 13. Τα σημεία 14 και 15 είναι πολύ γρήγορα, χωρίς προβλήματα και μπορούμε να τα κάνουμε αμέσως μετά, εάν υπάρχει χρόνος. Αλλιώς μπορούμε να τα περάσουμε σε μία επόμενη συνεδρίαση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άλπερτ Ντες, να ακούσουμε στη συνέχεια τον Τάσο, τον Νιώτη και μετά τους Κιώδης. Άλπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα σύντομα να παρουσιάσω πώς έχουν τα πράγματα, γιατί βασικά θέλω να ακούσω τη συζήτηση Ξέρετε την έκθεσή μου, την έχω καταθέσει, την έχετε διαβάσει και καλά. Όπως είπες, ε, Πάολο, 1267 στον αριθμό οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, αυτές που έμειναν δηλαδή, γιατί είχαν κατατεθεί και παραπάνω. Τις τροπολογίες αυτές, όπως ε, και πολλές άλλες, τις εκτίμησα και εδώ τις διάβασα το Σαββατοκύριακο. Βλέπετε πόσα, πόσες σελίδες ε, θα να σας πω στατιστικά 195 τροπολογίες ήταν για τα 16 σημεία της αιτιολογικής σκέψης. Μία τέτοια έκθεση είναι περιορισμένη και αν κάποια δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συμπεριλαμβάνονται, αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να έχει μία, ένα ορισμένο μέγεθος αυτή η έκθεση. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρονται οι μέλησες. Αυτό θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στις αιτιολογικές σκέψει, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου έκανε εντύπωση ότι έγιναν ε, για τις αιτιολογικές σκέψεις 195, γιατί παραγράφω παραγράφου ε, 1 έως 5. Είναι γενικά τα στοιχεία εδώ. Αναφέρεται η σταθερή χρηματοδότηση της αγροτική πολιτικής. 99 τροπολογίε κρατέθηκαν. Οι πιο πολλέ ε, τροπολογίε το περίμενα άλλωστε, αναφέρονται στα 14 σημεία για τις άμεσες πληρωμές. 326 τροπολογίες κατατέθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις συζητήσεις ε, κατά τις οποίες, ε, στις οποίες έκανα στην ομάδα μου, αλλά και σε άλλες ομάδες, αποκρισταλώνεται με σαφήνεια ότι μιλάμε για ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό στα ποσοστά ασφαλώς είναι πολύ και διαφορε... πολλές διαφορετικές οι απόψεις, πολύ διαφορετικές οι αλλά για τις πιο δίκαιες άμεσες πληρωμές μεταξύ των κρατών μελών, στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών, αυτό φυσικά μπορούμε να τσακωθούμε για το τι σημαίνει ακριβώς δίκαιη κατανομή, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να, θα πρέπει να βρούμε μια λύση για τις πιο δίκαιες άμεσες πληρωμές σε ό,τι αφορά τους πόρους και την περιβαλλοντική πολιτική. 7 σημεία, 143 τροπολογίες που κατατέθηκαν για τα 7 αυτά σημεία. Αν αφήσουμε κατά μέρο τις ακραίες ε, θέσεις, θεωρώ ότι και στο σημείο αυτό δεν απέχουμε τόσο πολύ και κατά τις επόμενες εβδομάδες θα καταφέρουμε να βρούμε συμβιβασμούς. Η τήρηση άλλων ε, υποχρεώσεων πέντε σημεία για τα οποία έλαβα 51 τροπολογίες και για το θέμα της, τροπο... της απλούστευσης. Δεν θέλουμε να καταστεί πιο περίπλοκη η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό συμφωνούμε μεταξύ των ομάδων. Δεν θα ανταποκριθούμε στο έργο μας αν δεν καταφέρουμε μετά το 2014 η γεωργία να έχει καταστεί πιο απλή. Οι γεωργοί πραγματικά δεν πρόκειται να δείξουν κατανόηση αν η όλη κατάσταση περιπλακεί περαιτέρω γραφειοκρατικά. Ήταν μια σημαντική απόφαση αυτή της ομάδας μου και είπαμε ότι με σαφήνεια, με σε κάθε περίπτωση ένα νέο σύστημα ε, με πληρωμών, κυρώσεων ελέγχων θα μας βρει αντίθετους. Θα πρέπει να περιορίσει τις σχετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε με την πολλαπλή συμμόρφωση είτε να συμπληρωθούν τα ήδη φυστάμενα μέσα μέσω του δεύτερου πυλώνα, όπου πολλά κράτη έχουν σημειώσει επιτυχία. Για τα 16 σημεία για τα μέσα της αγοράς πρόκυψε μία πρώτη επισκόπηση από την οποία καταδεικνύεται ότι υπάρχει ομοφωνία, συνένεση και ότι θα χρειαστεί να δίκτυο ασφάλειας και μετά το 2014. Κάτι άλλο που μου προκάλεσε έκπληξη είναι ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου Μόνο 160 τροπολογίες κατατέθηκαν. Σε εισαγωγικά το μόνο. Και σε κάποια σημεία μπορούμε απλά να αλλάξουμε κάποιες λέξεις. Αλλά γενικά υπάρχει ευρεία συνένεση ότι θέλουμε να συνεχίσει η θετική ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να διάσει η υπεθρός μας. και ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το εισόδημα στην Ήπεθρο, τα εισόδηματα στην Ήπεθρο. Και για το σημείο 57 καταδέθηκαν πολλές τροπολογίες. Ξέρω ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για την φορολογική πολιτική, αλλά πολλοί επιθυμούν να αναφερθεί μια υπόδειξη προς τα κράτη-μέλη ότι η φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ιδιαίτερη κατάσταση των γεωργών. Δεν θέλουμε να λάβουμε κάποια απόφαση, μπορούμε όμως τουλάχιστον να δώσουμε μια τέτοια υπόδειξη για τα κράτη-μέλη, για το τι επιθυμούν πολλοί αγρότες. Ελπίζω λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες να γίνουν διεξοδικότατες συζητήσεις. Προετοίμασα και κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις θα εργαστώ σκληρά προκειμένου να συνάψω συμβιβασμούς και με τις άλλες ομάδες για την έκθεση αυτή. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αν υπάρχει καλή θέληση, μπορούμε, θεωρώ, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καινούργια κατεύθυνση που πρέπει να πάρει μετά το 2014 η αγροτική πολιτική. Το αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτό. Όλοι θα πρέπει να αντιληφθούμε, άλλωστε ότι σε μια τέτοια σημαντική έκθεση, σε μια τόσο σημαντική απόφαση για το νέο προσανατολισμό της αγροτικής πολιτικής βρισκόμαστε σε πρώτη φάση σε διαδικασία συναπόφασης και θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου, αυτό ασφαλώς και θα επηρεάσει και το νομοθετικό ε, κείμενο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποφασίσουμε λοιπόν τι μπορούμε να υποστηρίξουμε και τι θα θέλαμε να τροποποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ωραία, ευχαριστούμε τον Άλμπερτ. Αν συμφωνείτε τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, Τάσο Νιώτη καταρχάς για να έχουμε και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα γίνονται και στη συνέχεια θα δώσω το, ρόλο στους, το λόγο στους κοιόδης οδητής. Παραγώ Τάσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για όλα όσα έχει κάνει για την έκθεση αυτή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προετοιμασία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναφέρθηκε ήδη με την παρέμβαση του Υπουργού υπάρχει ευρύτερη συνένεση όταν αφορά τους στόχους της ε, κοινή αγροτική πολιτική. Ευρύτερη συνένεση όχι μόνο από τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά και στις δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει κατά την προετοιμασία της ανακοίνωση και αυτή που γίνεται ε, κατά την προετοιμασία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να συζητηθούν, όπως ε, το επίπεδο του προπολογισμού, αλλά θεωρούμε ότι η συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μας επιτρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά εμάς, και θα είμαι πολύ σύντομος, υπάρχουν τρεις ευρύτεροι τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ιδέες μας προς το, παρα... παρόν. Καταρχάς να στοχεύουμε καλύτερα στην υποστήριξη το πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής και είναι πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής και στους δύο πυλώνες και τα θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας που θα βελτιώσουν την μελλοντική ευρωπαϊκή γεωργία. Όσον αφορά τώρα στο να επικεντρωθούμε καλύτερα στις ενισχύσεις. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στις ενισχύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι βασικό στοιχείο. Εάν υπάρχει αντίστοιχη οικονομική κατάσταση και αντίστοιχη κατάσταση όσον αφορά τον, ε, ε, στοιχείων που παραδίδονται δεν θα υπήρχε συζήτηση. Ο λόγο για τον οποίο γίνεται συζήτηση είναι γιατί θέλουμε να απομακρυνθούμε από ένα σύστημα που αντικατοπτρίζει το προηγούμενο επίπεδο ενίσχυση των παραδοσιακά επιστοριζόμενων τομέων προ ένα σύστημα το οποίο θα αντικατοπτρίζει καλύτερα αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Και για την υποστήριξη του βασικού εισοδήματο και για την υποστήριξη για τα δημόσια αγαθά. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο γίνονται συζητήσεις για το βαθμό της σύγκλησης. Τώρα, τη μεταβατική περίοδο επίσης, καθώς επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν με την κατανομή των ενισχύσεων στα κράτη-μέλη τα ίδια. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά, ε, διότι πρέπει να γίνει σωστή κατανομή όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και εντός των κρατών μελών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό το λεγόμενο πρασίνισμα. Εδώ υπάρχει ένας βαθμός ε, παράδοσης δημοσίων αγαθών, κυρίως ε, αγροτικών και περιβαλλοντικών αγαθών, ε, στο δεύτερο πυλώνα. Αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο της ευρωπαϊκής γεωγραφικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να περάσουμε σε ένα σύστημα όπου θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα συνδυάζουν κίνητρα για το 100% της αρρώσιμης έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχουν και κάποια επιπλέον μέτρα πολύ πιο στοχευμένα για το δεύτερο πυλώνα. Και τονίζω εδώ ότι τα μέτρα αυτά, επειδή ακριβώς πρέπει να ισχύουν για όλη την επικράτεια, θα πρέπει να είναι απλά και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση επιπλέον για τα κράτη-μέλη. Ορισμένες φορές μας επικρίνουν ότι εισαγάγουμε μέτρα που είναι πιο δαπανηρά για τους ε, γεωργούς. Ε, κάποιες άλλες φορές μας επικρίνουν γιατί πληρώνουμε χρήματα στους γεωργιούς για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Στην πράξη βιώνουμε σε μια κατάσταση όπου ακόμα και οι φυστάμενες πρακτικές που θεωρούνται βέλτιστες ε, κινδυνεύουν πλέον διότι αυξάνει πολύ το κόστος παραγωγής για τη γεωργία και επομένως ε, θα έχει πολύ σημασία πώς θα σχεδιαστούν εν τέλει αυτά τα μέτρα για το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα και πώς θα σχεδιαστούν με το δεύτερο πυλώνα. Όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα μέτρα αυτά, είναι σαφές ότι υπάρχει ε, δυνατότητα να κάνουμε τις ανάλογες προσαρμογές για αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προτεραιότητες που έχουν σχέση με την αλλαγή του κλίματος, με την πληροφόρηση και με την ε, απαραίτητη αναδιέρθυση της ευρωπαϊκής γεωργίας για να έχουμε αποτελέσματα. Αυτοί λοιπόν είναι οι βασικοί τρεις τομείς στους οποίους προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και προσβλέπουμε και στα αποτελέσματα της έκθεσής σας και της απόψης σας για να τις λάβουμε υπόψη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή Τάσο Χανιώτη. Να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση και να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης συζητητές. Ο Στεφάν Λεφόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Άκουσα μόλις και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και αναρωτιέμαι ε, περί τίνος η συζήτηση. Ποια είναι τα σημεία τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή προς τα πού βαδίζουμε, ποιο είναι το κείμενο που θέλουμε να εξαγάγουμε σε σχέση με την ανακοίνωση της Κομισιόν. Η ανακοίνωση ε, έχει διατυπώσει ένα κείμενο που βάζει ας πούμε τέσσερις μεγάλους στόχους στο θέμα της, ε, του πρασινίσματος και το ε, πρώτο πυλώνας. Ούτε λέξη. Τι επιλέγουμε πρώτο, δεύτερο, τι θέλουμε, πώς θα το πετύχουμε. Κανείς δεν συζητάει αυτά τα θέματα. Είχαμε πει κατά δεύτερο λόγο το θέμα του κοινωνικού μικρές εκμεταλλεύσεις, όρια, ενισχύσεων, συζήτηση νόμιμη. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα. Τρίτο σημείο για το θέμα της ρύθμισης. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη συμφωνία ότι θα υπάρχουν δίκτυα ασφάλειας. Ωραία. Αν έχουμε συμφωνήσει, τότε υπάρχουν αυτά τα δίκτυα τα ασφαλιστικά. Αλλά αν είναι αυτή η συζήτηση, ε, δεν χρειάζονται τρει ώρε. Υπάρχουν όμω πολιτικέ επιλογέ που πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ, εκ μέρου των σοσιαλιστών, λέω ότι οι 1200 τροπολογίε δεν είναι δικέ μα. Ε, προέρχεται από την οικογένεια του Albert Ντες. Εμείς στοχοθετήσαμε κάποιες τροπολογίες για να θέσουμε τα βασικά ερωτήματα. Τι θα κάνουμε για το πρασίνισμα αυτής της κοινωνικής της αγροτικής ε, πολιτικής είναι στον πρώτο ή στο δεύτερο πυλώνα. Έχουμε κάνει την επιλογή της διεύρυνσης των καλών γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα για να έχουμε μία ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική που να είναι βιώσιμη. Γιατί αν τα βάλουμε στο δεύτερο πυλώνα βούμε ε, να έχουμε μια ποικίλη περιβαλλοντική πολιτική. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την επιλογή και περιμένουμε μια απάντηση. Τι μας λένε τώρα, τι επιθυμούν να γίνει. Επίσης, όπως είπε ο συντονιστής ο τους προηγούμενους, κάναμε μια επιλογή ως προς τα επίπεδα των ορίων των ενισχύσεων. Έχουμε κάνει προτάσεις για το θέμα των μικρών εκμεταλλεύσεων και των ε, ε, και επίσης προτάσεις για το θέμα της ρύθμισης, ιδιαίτερα υπερασπιζόμενοι σταθερά και στεναρά τα θέματα που έχουν σχέση της οργανώσεις των αγροτών. Και τέλος για το θέμα το αγροτικό, είπα σε ένα κείμενο ε, κοινοβουλίου δεν μπορούμε να το δούμε μόνο ως προς το πώς θα χρηματοδοτηθούν και να συγχρηματοδοτηθούν οι ενισχύσεις. Έχουμε επίσης προτάσεις για να βάλουμε πολύ ουσία και νόημα σε αυτή τη θέση του Κοινοβουλίου. Ορίστε τι έχουμε επιτάπητος. Τώρα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε τους στόχους, όπως το κάναμε μόλις πριν από λίγο, με τον Υπουργό. Συμφωνούμε για τους στόχους. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, βιώσιμοι, αηφόροι και ταυτόχρονα να έχουμε επιστημιστική ασφάλεια για τους, όλους τους καταναλωτές. Τώρα, αυτά είπαμε όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα και εγώ δεν μπορώ να βλέπω να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση και να αφήσουμε στην Κομισιόν και το Συμβούλιο να αποφασίσουν ποιε είναι νομοθετικά, νομοθετικά μέτρα. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει τις ευθύνες Του με τους ε, συναδέλφους και τις ομάδες που το επιθυμούν θα πρέπει να ε, υποβάλουμε συμβαστικές τροπολογίες για να δώσουμε μια μεγαλύτερη ορατότητα και περιοπή ως Ευρωκοινοβούλιο προς όλους τους Ευρωπαίους αγρότες. αγρότες. Αυτό είναι το διακύβευμα και αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ Στεφάνο, George Λάιον και μετά ο Μάρτιν Χάουσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες των φιλελευθέρων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να γνωρίζουμε ότι το 55% των 1280 περίπου τροπολογιών που έχουμε είναι από την ίδια την ομάδα του Άλμπερτ. θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια κοινή θέση για όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά και κάποιοι μεταξύ μας. Η θέση που έχουμε εμείς και είχαμε εξ αρχής είναι ότι η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η δικαιοσύνη θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης και χρειαζόμαστε ένα απλό σύστημα, μία απλή κάπ για τους κανόνες, τους κανονισμούς και το πώς εφαρμόζονται και αυτό διέπει όλο το σκεπτικό της ομάδας μας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη κατανομή της χρηματοδότησης και αυτό φυσικά δεν είναι εύκολος στόχος. Και όπως είπε και ο Τάσος Χανιώτης, ο ίδιος ο στόχος δεν ε, επαρκεί. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε και αυτό συμπληρώνει και λίγο αυτά που είπε και ο Άλμπερτ ε, επί του θέματος δεχόμαστε το επιχείρημα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρηματοδότηση στον πυλώνα 1 και τη χρηματοδότηση στον πυλώνα 2, αλλά σαφώς δίνεται διαφορετικέ προτεραιότητε και επομένω για διαφορετικού στόχου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά κριτήρια για να ξέρουμε τι επίπεδο χρηματοδότηση θα έχουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη χρηματοδότηση και στους δύο πυλώνες, και στον 1 και στο 2, να ξέρουμε ότι αφορούν αρκετά διαφορετικές πτυχές και δεν μπορούμε απλώς να τα συγχωνεύσουμε και να πούμε ορίστε να τα ε, κάντε την κατανομή. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Όσον αφορά τώρα τις άμεσες ενισχύσεις, ε, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένες, θα πρέπει να ε, περάσουμε στο ίδιο σύστημα να την Ευρώπη και θα πρέπει να σταματήσει αυτό το ιστορικό σύστημα που χρησιμοποιούμε μέχρι το 2020 και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και κάποια μέτρα για το πρασίνισμα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα και αυτά αποτελούν βασικό στόχο κάθε φορά που εισάγονται μέτρα για το πρασίνισμα. Θέλουμε να έχουμε μέτρα τα οποία όχι μόνο θα βελτιώνουν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα αλλά και την οικονομική αποτελεσματικότητα και αποτελούν το βασικό για τους ε, ε, παραγωγούς και τους γεωργούς. Δεν θέλουμε να χαθεί η ευρωπαϊκή γεωργία επειδή θα είναι πιο πράσινες οι άμεσες ενισχύσεις. Συμφωνώ επίσης ε, με κάποια από τα στοιχεία που ανέφερε ο Άλμπερτ ένα νέο σύστημα συμμόρφωσης θα πρέπει να το απορρίψουμε ε, διότι θέλουμε να έχουμε μια πιο πράσινη ΚΑΠ και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα ταιριάζει με το παρόν σύστημα ε, ελέγχων και θα πρέπει να εφαρμόζονται πιο αυστηρά τα μέτρα κατά την άποψή μας. Κατά βάση θα πρέπει να στοχεύουμε κυρίως στους γεωργούς. Αυτό είναι το ουσιώδες. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, αυτό το έχουμε αναφέρει, θέλουμε να έχουμε πράσινη ανάπτυξη, καινοτομία, περιφερειακά μέτρα για το περιβάλλον και οποιοδήποτε πιο πράσινη άμεση ανίσχυση θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ε, αλλαγή του κλίματος και τη βιωσιμότητα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ο καθένας τοπικά, θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα για τα ανώτατα όρια δεν συμφωνούμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω το εφιστάμενο σύστημα, το σύστημα τώρα μικρής κλίμακας. Εμείς είμαστε υπέρ της πραγματικής απλούστευσης του συστήματος. Δεν θέλουμε να ε, τιμωρήσουμε τους μικρούς γεωργίους ανά την Ευρώπη, τα μέτρα αυτά θα, για τους μικρούς γεωργούς θα πρέπει να είναι προαιρετικά. Επίσης θεωρούμε ότι θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ένα κατεπήγον δίκτυο ασφαλείας για να αντιμετωπίσουμε κρίση. Εμείς ως ομάδα ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε με άλλες πολιτικές ομάδες για να υπάρχει ε, ένα συμβιβασμός, ε, συμβαστικές προτάσεις που θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη ΚΑΠ. Αλλιώς νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θα μας λάβουν σοβαρά υπόψη και ελοχεύει και ο κίνδυνος να μην συμφωνήσουμε και να μην προκύψουν κάποια στεναρά μηνύματα από την έκθεση αυτή, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ε, για το νομοθετικό πακέτο. Βέβαια, για να ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να φτάσουμε στι αρχέ του επομένου χρόνου. Έτσι έχουν τα πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συνεργαστώ με του υπολείπου για να έχουμε μια ισχυρότερη ΚΑΠ, γιατί αυτό άλλωστε είναι και ο στόχο μα. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι για να έχουμε περισσότερη πολιτική βαρύτητα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάρτιν Χάουσλινγκ τώρα. Συνάδελφοι, αναρωτιόμαστε γιατί συζητάμε σήμερα ένα σημείο όπου όλοι διαβεβαιώνουμε ένα τον άλλον ότι έχουμε κοινούς στόχου και τελικά καταλήγουμε να λέμε αυτά που έχουμε πει πέντε φορές. Νομίζω ότι πολύ απλά βρισκόμαστε σε ένα σημείο ε, που θα ήθελα να συζητήσουμε συμβιβαστικές ε, προτάσεις από πλευράς του εισηγητή. Το βασικό πρόβλημα της έκθεσης είναι ότι η πολιτική οικογένεια, του ΕΛΚ μας δυσκολεύει. Γιατί δεν ξέρει σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί. Νομίζω ότι όταν συζητάμε για σεμιβασμούς θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε αυτά που μας έχει δώσει, μας έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι στην πρώτη συζήτηση συμφωνήσαμε ότι θέλαμε να συμφωνήσουμε επί της ουσίας, ε, επί της πρότασης της μεταρρύθμισης. Τώρα το θέμα είναι πόσο πρόθυμοι είμαστε όλοι να συνάψουμε συμβιβασμού για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε μια δυνατή μια ισχυρή τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Και όχι να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία τελικά να μην λέει τίποτα, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα μας πάρουν στο σοβαρά ως Κοινοβούλιο. Δεν θα σας παρουσιάσω όλες μας τις τροπολογίες από πλευρά των Πρασίνων θεωρώ ότι θα πρέπει να καταστήσουμε διακριτό το Κοινοβούλιο να εργαστούμε για μια μεταρρύθμιση και να μην περιοριστούμε μόνο στην μείωση της γραφειοκρατίας, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε καλές πιθανότητες να πετύχουμε. Δεν μπορεί η μείωση της γραφειοκρατίας να αποτελεί τον τίτλο μιας αγροτικής μεταρρύθμισης από πλευρά του Κοινοβουλίου άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Και βασικά το θέμα είναι η συμβατότητα με θέματα περιβάλλοντος και με την πολιτική το 2020. Ωραία, ας περάσουμε τώρα στις λοιπές παρεμβάσεις. Σας παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο λακωνικοί. Ιδάλλως θα πρέπει να περιορίσουμε κατά πολύ το πολύ σημαντικό εργαστήριο που έχουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση είναι πολύ περίπλοκη και δύσκολη. Ο αριθμός και μόνο των τροπολογιών υποδεικνύει το πόσο περίπλοκη είναι αυτή η έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την έκθεση υπάρχουν πολλαπλές προσπάθειες αντικατάστασης των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν. Υπάρχει ένα εγχείρημα να αλλάξουμε την πορεία των προτάσεων, διότι αυτές οι νομοθετικές προτάσεις δεν θα πρέπει να προέρχονται από τη δική μας Επιτροπή, αλλά από την Κομισιόν. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Η προτινόμενη μεταρρύθμιση είναι πολύ ρηχή. Στην πραγματικότητα είχε ανακοινωθεί ως κάτι το ρηξικέλευθο, αλλά σε τελευταία ανάλυση φαίνεται κάτι το πολύ συντηρητικό να προκύπτει. Περιγράφεται ως ανοιχτή, σύγχρονη και ρηξικέλευθη. είναι γι' αυτό που υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί. Δεν αναφέρονται αρκετά για τα μέσα της αγοράς, για τη σταθερότητα της αγοράς. Και τα μέσα της αγοράς και τα εργαλεία είναι πιο σημαντικά από το πώς υλοποιούνται οι πληρωμές. Διότι οι αγρότες ε, θέλουν να βγάλουν ε, λεφτά από την παρουσία τους στις αγορές και χρειάζεται σταθερότητα. Το πρασίνισμα της πολιτικής ακούγεται ωραίο, ακούγεται καλό. Η κοινή γνώμη το προσλαμβάνει με θετικότητα. Έχουμε ήδη υψηλά πρότυπα. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, ας την κάνουμε ακόμη πιο πράσινη και προσανατολισμένη περιβαλλοντικά. Έχουμε επίγνωση της ανάγκης να ε, εξασφαλίσουμε την, ασφάλεια, την επιστημική ασφάλεια, αλλά ας μην πάμε πολύ μακριά. Ας θυμηθούμε τις συνόδους κορυφής ε, για τις κλιματικές ε, αλλαγές. Ήταν φιάσκο και οι δύο σύνοδοι κορυφής. Ας μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στη Γεωργία. Βέβαια, αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στήριξης. Αλλά η γεωργία χρειάζεται διαφορετικά επίπεδα στήριξη. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν μπορούμε να δούμε την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μόνο από περιβαλλοντική άποψη. Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Γι' αυτό θα πρέπει να αντισταθμίσουμε ε, εκείνες τις χώρες που ε, χρειάζονται ισχυρότερη ανάπτυξη της υπαίθρου διότι έχουν μείνει πιο πίσω από τις άλλες. Θα πρέπει να πετύχουμε συνένεση και ε, έχουμε καλή τύχη σε όλους σε αυτό το στόχο. Ο κύριος Άκνιο και μετά ο Σέριτζιο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εξή. Αναφερθήκατε στους τρεις ε, τομείς, ε, στους οποίους επικεντρωνόσαστε πρασίνισμα, καλύτερη επικέντρωση και καινοτομία, αν κατάλαβα καλά. Και εκεί αρχίσατε να μας λέτε για την αλλαγή του κλίματος. Τα μέλη της Επιτροπής θα γνωρίζουν την άποψή μου επί του θέματος, αλλά οι περισσότεροι εδώ στην Επιτροπή μας θεωρούν ότι οι δραστηριότητες των γεωργών θα υπογαρεύουν τον καιρό, ενώ εγώ θεωρώ ότι ο καιρό υπαγορεύει αυτά που κάνουμε, έτσι πίστευαν οι Γεωργοί. Τι θα κάνετε με αυτό, τι θα ζητήσετε από του Γεωργούς να κάνουν για να αλλάξουν το κλίμα. Ακούσαμε πριν από ένα χρόνο εδώ μια παρουσίαση όπου είπατε ότι θα πρέπει να θάβετε το διοξίδιο του άνθρακα και να μην έχουμε αέρια. Βέβαια αυτά θα αλλάξουν πολύ. Θα πρέπει όμως να μας πείτε τι περιμένετε να κάνουν οι Γεωργοί για να αλλάξουν το κλίμα και πόσο θα κοστίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο Σέργιο Γουτιέρης και μετά ο κύριος Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, επί της εκθέσεως αυτής, το πιο σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί και τον κοινό παρανεμαστή σε όλα όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να έχουμε μια δίκαιη ΚΑΠ. Τι σημαίνει δίκαιη ΚΑΠ να είναι παρκής, ισχυρή, εντάξει, δεκτό, αλλά δίκαιη σημαίνει να έχουμε αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς και να μπορούν όλοι ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη τους δραστηριότητα και από το πώς αναπτύσσεται να διεξάγουν την εργασία τους. Και νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποια πράγματα σαφώς για αυτό το στόχο. Καταρχάς, άμεσες ενισχύσεις και διαχείριση των αγορών. Ακούσαμε ότι είναι φιλόδοξη η αγορά αυτή και ε, χρηματοδοτείται επαρκώς και εμεί ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποστείλουμε στεναρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να χαθούν κάποια πράγματα ούτε στις άμεσες ενισχύσεις ούτε στα υπόλοιπα. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στο ολοένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον και αν θέλουμε να προσαρμοστούμε και στη στρατηγική 2020 το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κοινό παρονομαστή για τη στρατηγική μας. Κάποιες προτεραιότητες. Καταρχάς να επαναλάβω τη σημασία των μεταβατικών περιόδων. Από να είναι ομαλή η μετάβαση για να μπορέσουμε να περάσουμε από την ε, πολιτική για την ΚΑΠ του 2013 στην πολιτική μέχρι το 2020. Μία πολιτική που θα σχετίζεται και με την απασχόληση γιατί για να είναι δίκαιη η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι και κοινωνική ΚΑΠ και επίσης πέραν της ενίσχυσης ε, των μέσων της αγοράς ε, κυρίως όσον αφορά το, τις ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις τιμές παρέμβασης. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το διαπιστώσαμε και με την ε, ε, κρίση του ελαιολάδου όπου είχαμε τιμές πολύ χαμηλότερες και εκεί δημιουργήθηκαν επιπλοκές για να μπορέσει κάποιος ε, να λάβει και τις ενισχύσεις. Μία δίκαιη ΚΑΠ επίσης θα πρέπει να δίνει και δυνατότητα ε, διαπραγμάτευσης στους ε, γεωργούς και στους παραγωγούς. Θα πρέπει όπως ε, περιλάβαμε μέτρα στα γαλακτοκομικό τομέα να περιλάβουμε και σε ολόκληρη την ΚΑΠ και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί συντελεστές στην ερμηνεία των εθνικών κανόνων διότι είναι πολύ διαφοροποιημένη η κατάσταση. Τέλος, όσον αφορά τις ε, γεωργικές εκτάσεις ε, είναι πολύ σημαντικά κατά την άποψή μας και ορισμένες φορές δεν τις αναφέρουμε παρκώς. Δύο ιδέες θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ για να καταστήσω κάτι σαφές. Καταρχάς θα πρέπει να παραμείνουν αυτά τα θέματα με τις γεωργικές εκτάσεις ε, στις χώρες που τα έχουμε χρησιμοποιήσει όπως είναι η Ισπανία και να κάνουμε και ένα βήμα περισσότερο σας Έχουμε εγγυήσει, για παράδειγμα, σαν αυτέ του Καναδά, που θα μπορούσαν να είναι απόλυτα συμβατέ με το πράσινο κουτί του ΠΟΕ και που θα μα επιτρέπουν, επειδή ακριβώ είναι συμβατά με του κανόνε του ΠΟΕ, να έχουμε μέχρι και το 60% ανάκτηση των απολειών και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αγορά. Θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ σημαντικέ και θα μπορούσαμε να τι συμπεριλάβουμε στην έκθεση και είμαι πεπισμένο ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρξει συνεννόηση επί του θέματο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Παπαστάμκος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, επειδή ακούστηκαν οι τροπολογίες πολλές που κατέθεσαν, ε, καταθέσαμε οι συνάδελφοι του ΕΛΚ, θέλω να πω ότι εμείς τιμούμε το έργο του κυρίου Ντές, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι και το Λαϊκό Κόμμα είναι ένα πολύ πλουραλιστικά ε, δομημένο κόμμα, εξού και αυτές, ο μεγάλος αριθμός συνεισφορών ε, μέσω το, των τροπολογιών. Εν το, το, το ζητούμενο είναι, και εγώ συμφωνώ με, με της συναδέλφους, το ζητούμενο είναι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κωδικοποιήσουμε το δικό μας πολιτικό μήνυμα κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και να συμπέσουν οι απόψεις μεταξύ περισσότερων ομάδων, εδώ κοινοβουλευτικών, σε 5, 10, 15 σημεία. Νομίζω τότε και το μήνυμά μας ε, θα είναι ηχηρό. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις, διαφορετικές αναγνώσεις προς το μέλλον της ΚΑΠ. Κάποιο είπε, «Ε, δεν είναι μεγάλη αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα και χρησιμοποίησα και παλαιότερα τη λέξη, όχι reform, αλλά evolution της ΚΑΠ. Ε, και εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί έχουμε ένα άλλο πρότυπο γεωργία στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Δεν έχουμε γεωκτήμονε με τεράστιε εκτάσει. Έχουμε μικρού καλλιεργητέ, κύριε Πρόεδρε. Και γι' αυτό και υποστηρίζω, παραδείγματο χάρη, ότι πρέπει να μπει οροφή στι ε, άμεσε ενισχύσει. Σέβομαι από την άλλη πλευρά συναδέλφου που αντιτίθενται στη θέση οροφή. Όμω δεν είναι το ίδιο ένα μεγάλο γεωκτήμονα, ένα που κατέχει αρκετέ δεκάδε εκταρίων και καλλιεργεί, με αυτόν ο οποίο ε, ο μέσο όρο γεωργική εκμετάλλευση είναι δύο ε, εκτάρια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επομένω και την ποικιλομορφία των καταστάσεων. Ε, τι θα πει δικαιότερη κατανομή. Ε, ακούω συνέχεια δικαιότερη κατανομή, δικαιότερη κατανομή. Να πάρουμε υπόψη μας το κριτήριο των δικαιούχων. Όχι το κριτήριο των εκταρίων. Λέω και μπορώ να το, ε, να το αντικειμενικοποιήσω αυτό που λέω. Βεβαίως από την άλλη δεν θέλω ε, να, να μακρηγορήσω. Ε, ακούω συνέχεια το πρασίνισμα. Βεβαίως το πρασίνισμα το χρειαζόμαστε αλλά κύριε Πρόεδρε, πρασίνισμα στην παγκόσμια κλίμακα. Το Η οικολογία, μάλλον η διατήρηση των θεμελίων της ζωής, δεν έχει μία μόνο σήμαντη ευαισθησία και δεν αφορά ένα τομέα ή μία παράταξη ή μία αντίληψη. Έχει, είναι, η διατήρηση των θεμελίων της ζωής είναι μία οικουμενική εντολή. Και γιατί έχει πλημμυρίσει η ευρωπαϊκή αγορά από προϊόντα τρίτων χωρών που δεν έχουν καθόλου ε, πρασίνισμα ή ελάχιστο πρασίνισμα. Αυτό δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διάσταση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια εμπορική κλίμακα. Ξέρω ότι πουλάει και συγχωρήστε μου τη λέξη ε, το, το πρασίνισμα, το πρασίνισμα, το πρασίνισμα γι' αυτό έχει εμπλουτίσει και τη ρητορική ε, και της Κομισιόν και των Επιτρόπων. Βλέπουμε εδώ έρχονται, παρελάβουν οι Επίτροποι αρμόδιοι στην αρμόδιοι και μιλούν για το, πρισίνι, το πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν ακούω κύριε Πρόεδρε από την Κομισιόν να μας λέει κάτι για το πρασίνισμα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες βιομηχανίες φυτοφαρμάκων, τις μεγάλες βιομηχανίες λιπασμάτων, τη χρήση αυτών των μέσων ε, σε ό,τι αφορά τη γεωργική παραγωγή. Και επειδή ακούγεται, εγώ αν εξαιρέσω τους υδάτινους πόρου, θέλω να πω για τη χώρα μου ότι είναι η πρώτη ή η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με δεσμευμένες εκτάσεις στο πρόγραμμα Natura. Δηλαδή εξορισμού είμαστε μια φιλοπεριβαλλοντική χώρα όπως θέλουμε να μετρούμε με αυτά τα κριτήρια της, ε, της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E Ευχαριστώ Γιώργο. Και τώρα η κυρία εραντ Καρσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, διαπράττουμε το ίδιο σφάλμα που διαπράττουμε πάντα. Ε, κάνουμε όλες τις αποφάσεις ε, πριν ολοκληρωθεί ο γύρος ε, του ΠΟΕ. Οτιδήποτε αποφασίσουμε για το πρασίνισμα θα μας τα φέρουν ανάποδα αν θέλετε πριν ε, ολοκληρωθεί ο γύρος. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε στις διαπραγματεύσεις και όταν θα γνωρίσουμε τι συμφωνείτε εκεί να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, γιατί αλλιώς θα κάνουμε διπλή προσπάθεια όπως κάνουμε συνήθως. Και αν συγκριθούμε με τα άλλα συμβαλόμενα μέσα διαπράγματευση, ε, θα ξέρετε ότι οι τρίτες χώρες δεν θέλουν ούτε να ακούσουν τα θέματα αυτά και οι Ηνωμένε Πολιτείε προστατεύουν ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή του ε, τομέα, ενώ εμεί τον αποδυναμώνουμε. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υπόθεση αυτή. Μιλήσαμε για την πολιτική βαρύτητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μέσω αυτών των εκθέσεων ότι ε, έχει μια συνοχή Έχουμε την έκθεση Λάγιο, την έκθεση Νταντάν, ακόμα και την έκθεση του κυρίου Μποβέ, την οποία υποστήριξε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή μας έδειξε ότι έχει μία σαφή γραμμή που θέλει να προστατεύει τον πρωτογενή τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή η εικόνα της συνοχής θα πρέπει να χαθεί. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να βοηθάμε και να χαθεί ο, διαχωριστεί ο πρώτος πυλών από το δεύτερο και να θεωρήσουμε ότι είναι ανεξάρτητα τα δύο πράγματα στη διαπραγμάτευση για τις δημοσιονομικές προοπτικές και να χαθούν όλα όσα κατάφερε να ε, πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενες εκθέσεις. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, και να υπάρχει αμοιβαιότητα και να είμαστε σοβαροί με τον ΠΟΕ. Όλα όσα προτείνουμε συστηματικά είναι όλα όσα έχουμε συμπεριλάβει εμείς στις τροπολογίες μας στην έκθεση και αυτό είναι ε, το μεγάλο τμήμα των τροπολογιών που παρουσιάστηκαν. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες θέλουν να βάλουν την έκθεση προς τη σωστή κατεύθυνση και εγώ λοιπόν θα ήθελα να υποστηρίξω ε, τις συμβαστικές τροπολογίες που παρουσίασαν κάποιοι συνάδελφοι από το ΕΛΚ. Κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Εγώ νομίζω ότι εμείς το ΕΛΚ ε, πλησιάζουμε στη συνένεση. Ε, συμφωνούμε περίπου με αυτά που συνάδε, ε, παρουσίασε ο συνάδελφος Μαριναϊσκού και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μία ισορροπία, μία έκθεση που θα υποστηρίζει την πρωτογενή παραγωγή και θα έχει και το 90% του υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πάντα αυτό συμβαίνει, διότι πάντα εργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό ο γύρο τραπέζη. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω από τον Τάσο Χανιώτη αν θέλει να παρέμβει. Αν δεν θέλετε να παρέμβετε, θα δώσω και πάλι το λόγο στον Άλμπερτ Τέσ και κατόπιν. Έχετε το... Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ο Τάσο Χανιώτη και μετά θα ολοκληρώσει ο Άλμπερτ Ντέσ. Σύντομα. Πολύ σύντομα, ε, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς δεν θα πούμε στους ε, αγρότες πώ να επηρεάσουν τον καιρό, αλλά πώς θα ανταποκριθούν στις αλλαγέ στις καιρικέ. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε συμφωνήσει και μου φαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται. Υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ του γνώσης που έχουμε για την αλλαγή του κλίματος και της ανάγκης προσαρμογής της γεωργίας και τα ερωτήματα που μας θέτουν οι αγρότες επιτόπου, ε, όταν μιλάμε για καινοτομία, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, αναπτύσσοντας συστήματα, συνδέοντας τις νέες επιστημονικές γνώσεις με τα ισχύοντα γεωργικά συστήματα. Και αυτό που προσπαθούμε να διευκρινίσουμε. Είναι σαφές όμως ότι η γεωργία ε, πολλά έχει κληθεί να κάνει σε ό,τι αφορά την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά θα κληθεί να κάνει και στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ιδέες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ Τάσο. Ο Άλμπερτ για να με εξαγάγει συμπεράσματα από τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε έχω κάποιες παρατηρήσεις και μπορώ να διαβάσω κάποια από τα στοιχεία αν έχουμε χρόνο. Έχω και κάποιες ε, συμβιβαστικέ να παρουσιάσω αν θέλετε, αλλά αν μου ασκείτε κριτική για την κατάθεση τροπολογιών από την ομάδα μου, ε, τι να πω. Δεν εύχομαι σε εισηγητές να έχουν τόσο ισχυρή ομάδα. Μια τόσο μεγάλη ομάδα από μέλη 26 χωρών είναι τόσο μεγάλη ομάδα μου όσο καμία άλλη ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις είναι κάτι που θα πρέπει να αποδεχτούμε. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχει ε, ποικιλομορφία ε, στην ομάδα μου, αλλά αυτό να μην απογοητεύει τις άλλες ομάδες. Θα βρούμε καλές συμβαστικέ ε, συμβαστικές προτάσεις ε, στην ομάδα μου. Προς τα που οδεύουμε να σας διαβάσω ένα σύντομο κείμενο, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Πέτυχα ένα συμβιβασμό στην ομάδα μας για το σημείο 9, ότι ζητά την σωστή κατανομή των μέσων μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των αγροτών στο εσωτερικό των ε, κρατών μελών και αναφέρουμε ότι θα πρέπει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή των πληρωμών αυτών για να βοηθήσουμε την παραγωγή των αγροτών ως κεντρικό στόχο και τάσεται υπέρ της συμπερίληψης συγκεκριμένων όρων πλαισίου στα κράτη-μέλη. Απορρίπτει ένα σύστημα καταποκοπήν πληρωμής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η συμβιβαστική πρόταση της ομάδας μου και μπορούμε να συζητήσουμε με τις άλλες ομάδες κατά πόσο συμφωνούμε με μια τέτοια πρόταση ή κατά πόσο υπάρχουν επιθυμίες να αλλάξει αυτή η συμβιβαστική πρόταση. Θα έχουμε χρόνο τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες και θα χρησιμοποιήσω το χρόνο αυτό για να κοιτάξω τα θέματα αυτά και να τα συζητήσω με τις διάφορες ομάδες. Ε, ο George Lyon μίλησε για το μεγάλο ποσοστό τροπολογιών από την ομάδα μου. Χαίρομαι που η ομάδα μου έχει ασχοληθεί τόσο εντατικά με το θέμα αυτό. Και να σας πω και ότι αν ε, είχα γράψει διαφορετικά την έκθεση αυτή και πάλι θα υπήρχαν πολλές τροπολογίες, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο που επικρατεί σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Να απαντήσει στον κύριο Χόισλινγκ, ο οποίος ε, είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε διάθεση και προθυμία για συμβιβασμό. Εγώ από πλευρά μου πάντα έλεγα ότι είμαι διαδεθειμένος να συμφωνήσω με λογικά πράγματα, αλλά αν και ο Χόισλινγκ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου μιλάνε μόνο για screening στη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής, συμφωνώ με την κυρία Έραντς. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε εδώ πράσινα κριτήρια χωρίς να ξέρουμε τι θα προκύψει από τον ΠΟΕ, τι θα προκύψει από τις διμερείς συμφωνίες με το Μερκοσούρ, με τον Καναδά. γιατί θα προκύψουν νέες πραγματικότητες και σήμερα δεν ξέρουμε πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό ξέρουμε ακόμα και εδώ αποφασίστηκε μια συμβιβαστική θέση της ομάδας μας για το άρθρο 23. Θεωρούμε ότι τα μέσα τα οποία θα δαπανηθούν για το πρασίνισμα θα πρέπει να εξαρτώνται από το σύνολο του προϋπολογισμού καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε πώς αυτή η υπερβραδική πτυχή μπορεί να χρηματοδοτηθεί, νομίζω ότι πρόκειται για μια πρόταση συμβιβαστική. Ποιος μπορεί να είναι αντίθετος με μια τέτοια προσέγγιση. Και να σας πω ότι αν νομίζετε ότι 80% ευρώ στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να αντικατασταθούν από πράσινους όρους Κοιτάξτε, αν ε, θεωρούμε ότι θα φορτωθεί κάποιος γεωργός 120 ευρώ κόστος για να συμμορφωθεί με τους όρους που απαιτούνται για να πάρει 80 ευρώ πληρωμή, τι νόημα έχει. Το, οι πράσινοι όροι σημαίνουν μείωση του κέρδους. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όποιοι με γνωρίζουν θα ξέρουν ότι είμαι υπέρ λογικών όρων. Όπου υπάρχουν ελλείμματα στην Ευρώπη για την περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να δράσουμε, να επέμβουμε. Αν όμως κράτη-μέλη ξοδεύουν ήδη 40% για την προστασία του περιβάλλοντος, τι θα έρθουν να πω στα κράτη-μέλη αυτά να προσθέσουν 10% περαιτέρω, ενώ υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν αφιερώνουν καν 5% για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ. Σικέρσκι επίσης ε, αναφέρθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής, χωρίς ε, να ασκήσω κριτική σε εγκαθνέναν, γιατί ξέρω ότι και στην Επιτροπή υπάρχουν άλλα συμφέροντα, να φέρω και τον Επιτροπό Εμπορίου για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι τόσο λεπτομερής για να μπορέσουμε να δούμε πώς αποτυπώνεται το μέλλον της αγροτικής πολιτικής. Ο συνάδελφος Αγνιό μίλησε για την αλλαγή του κλίματος. Θεωρώ και εγώ ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα ήθελα αριθμητικά στοιχεία για το ποσοστό της ε, συμβολής της ε, γεωργίας. Δεν νομίζω ότι τα ποσοστά είναι τόσο σημαντικά σε ό,τι αφορά τη δίκαιη κατανομή τώρα. Το είπε και ο συνάδελφος, το πρόβλημα αυτό ανακύπτει σε κάθε κείμενο, σε κάθε έκθεση. Τι σημαίνει δικαιοσύνη. Στο άρθρο 9 που σας διάβασα προσπάθησα να βρω μια δίκαιη λύση. Και στα άλλα άρθρα επιμένω να υπάρχουν σωστές μεταβατικές περίοδοι. Δεν είναι δυνατόν το 2014 να υπάρξει μια δραστική αλλαγή και όλοι οι γεωργοί να βρεθούν σε μια εκβάθρον διαφορετική κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνη, να δούμε τι θα αλλάξει στην επόμενη αγροτική περίοδο και να υπάρχουν οι σωστές μεταβατικές περίοδοι. Αναφέρθηκαν τα θέματα για την ασφάλιση του κλίματος. Αναφέρεται στην έκθεσή μου αυτό, ότι είναι θέμα των κρατών μελών. Θα πρέπει όμως να δίνουμε από ευρωπαϊκό επίπεδο τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα συστήματα αυτά. Στη Γερμανία δεν ακούω πολλά δεν υπάρχει μεγάλη επιθυμία για ένα τέτοιο σύστημα και σε αυτό το σημείο λοιπόν διαφέρουν σημαντικά τα 27 κράτη-μέλη. Ο κ. Παπαστάμκος αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να προσέξουμε για το ποιες διαφορές υπάρχουν στην Ευρώπη μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών και ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Το έγραψα ρετά στην έκθεση το θέμα των μικρών χωρών, των μικρών αγροτών. είναι τόσο σημαντικό στα 27 κράτη-μέλη που δεν μπορούμε από την, ε, στις Βρυξέλλες να ορίσουμε τι θα πρέπει να ισχύει για τους μικρούς αγρότες. Όχι, εμείς μόνο ένα πλαίσιο μπορούμε να δώσουμε. Για την κυρία Έραντς απάντησα. Τον κύριο Έραντς. Αν ε, με κατηγορείτε ότι η όλη συζήτηση περιστρέφεται μόνο γύρω από τη μείωση της γραφειοκρατίας, έχετε άδικο. Όχι, στο επίκεντρο είναι τα περιβαλλοντικά μέτρα. Εγώ επισκέφθηκα πολλές αγροτικές περιοχές, το είπε ο κ. που πουθενά δεν είδα πιο βιώσιμη γεωργία από ό,τι σε εμάς στην Ευρώπη. και είμαι πρόθυμος να συμπεριληφθούν και κάποια στοιχεία για το τοπίο. Νομίζω ότι μπορούμε να το εντάξουμε αυτό στον πρώτο πυλώνα. Δεν ενδιαφέρουν πολύ οι απόψεις μας και αν υπομονώ να ακούσω και τις μελλοντικέ συζητήσεις είμαι απόλυτα βέβαιος, επειδή ξέρω αυτή την Επιτροπή, ότι από πλευράς στόχων κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε τα πολλά παρακλάδια τα οποία ανοίγονται μπροστά μας να τα συνενώσουμε σε μια βασική οδό, την οποία και να ακολουθήσουμε η προσπάθεια που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε ευχαριστώ και εσένα, Άλμπαρτ, και όλου του και όλους Είμαι βέβαιο ότι εν τέλει θα βρούμε μια κατεύθυνση που θα αποτελεί και σημείο συνάντηση όλων των ευαισθησιών. Να περάσουμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη, διότι έχουμε τώρα την παρουσίαση τη μελέτη «Ποια εργαλεία για την κοινή γεωργική πολιτική για την υποστήριξη τη παροχή δημοσίων αγαθών». Τα σημεία 15 και 16 νομίζω ότι μπορούμε να τα αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας, ώστε να νιώσουμε λίγο πιο ελεύθεροι, Δεν, να μην υπάρχει κάτι κατεπήγον και να επικεντρωθούμε σε αυτή την τόσο σημαντική μελέτη. Καταρχάς, να καλωσορίσω στα μέλη της ε, ομάδας, τους εμπειρογνώμονες που είναι εδώ για να παρουσιάσουν τη μελέτη, τους κυρίους David Baldock, ε, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική, τον ε, πρέσβη Κοράντο Πίρτσιο Μπίρολη, τον οποίο έχουμε ακούσει επανειλημμένος εδώ στην Επιτροπή και που όπως γνωρίζετε είναι ο αντιπρόεδρος ε, του Ιδρύματος ΡΑΙΣ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλντοκ για να μας παρουσιάσει τη μελέτη και στη συνέχεια θα είναι στη διάθεσή σας και οι δύο μιλητές για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Όποιος δεν ενδιαφέρεται για τη μελέτη μπορεί να αποχωρήσει. Ελπίζω οι συνάδελφοι Ευρωβουλευτές να παραμείνουν στις θέσεις τους και να δώσω το λόγο στον Ντέιβιτ. Παρακαλώ, Ντέιβιτ. Thank you very much, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε τα βρήματα της μελέτης μας. Εδώ εκπροσωπώ μια ομάδα που περιλαμβάνει το Ίδρυμα και την ΕΝΕΑ στην Ιταλία και VTI στην Γερμανία. Και θα πρέπει να πω ότι η μελέτη δεν έχει περατωθεί πλήρως και προσβλέπουμε στις αντιδράσεις των μελών της Επιτροπής σήμερα θα περάσω στα πετάχτα τη μελέτη. Είμαι βέβαιος ότι έχετε δει αντίτυπο των ε, διαφανειών. Ίσως να θέλετε να θέσετε συγκεκριμένα ερωτήματα σε συγκεκριμένα θέματα. Η Επιτροπή μας έχει ζητήσει να ασχοληθούμε με ορισμένα θέματα. Πρώτον, ποια είναι τα δημόσια αγαθά που σχετίζονται με τη γεωργία στην Ευρώπη ποιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε, σε ποιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε ε, ως προς την ΚΑΠ, τι πολιτικές έχουμε, τι πολιτικές μπορεί να έχουμε μελλοντικά. Και θα προσπαθήσω συγκεκριμένα να ε, ασχοληθώ με το τελευταίο ζήτημα που είναι πιο συναφές στη συζήτηση που είχαμε, δηλαδή ποια θέλουμε να μελετήσουμε στο μέλλον. Πρώτον λοιπόν, ποια είναι τα δημοσιαγαθά που σχετίζονται με τη γεωργία και την δασονομία, δεν θα ασχοληθώ με τη δασονομία για να πλουστεύσω τα πράγματα και να κάνω την παρουσίαση πιο εύκολη. Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε το θέμα ότι ε, το κυριότερα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά είναι η βιοπικιλότητα της αγροτικής γης, ε, τα γεωργικά τοπία, ψηλή ποιότητα υδάτων, αέρα και εδαφών, σταθερότητα κλίματος, εδώ μιλάμε και για την μείωση των εκπομπών, αλλά και για την δέσμευση του άνθρακα ε, και την ανθεκτικότητα στις φωτιές και τις πλημμύρες. Υπάρχουν επίσης άλλα πολύ σημαντικά δημόσια αγαθά που δεν είναι περιβαλλοντική φύσεως. Υπάρχουν κάποια κοινωνικά και πολιτιστικά και τα συνοψίζουμε με την ορολογία αγροτική ζωτικότητα. Είναι έχει να κάνει με την ζωτικότητα των αγροτικών πληθυσμών και κοινοτήτων. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται με την γεωργία, σε άλλα μέρη της Ευρώπης η σχέση με την γεωργία δεν είναι τόσο ισχυρή. Η ε, ζωτικότητα είναι θέμα που αφορά όλες τις περιοχές. Έχουμε επίσης την ε, ορθή μεταχείριση των ζώων, εκτροφής και υπάρχει και το θέμα της επισυστιστικής ασφάλειας τροφοδοσία τροφίμων και η επισητιστική ασφάλεια, διατήρηση της δυνατότητας ε, του εδάφους και άλλων πόρων και δεξιοτήτων για την παραγωγή τροφίμων στο μέλλον. Αυτά είναι τα δημόσια αγαθά που σχετίζονται με τη γεωργία στην Ευρώπη. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αν είμαστε σε θέση να έχουμε πολιτικές που αποδίδουν περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, μπορούμε να έχουμε και κάποια κοινωνικά και πολιτιστικά δημόσια αγαθά λόγω ε, των σχέσεων με τον τουρισμό, την αναψυχή, επίσης ε, σε σχέση με την απασχόληση στις εκμεταλλεύσεις, εκτός εκμεταλλεύσεων, προσθέτουμε υψηλή αξία σε προϊόντα αγροτικά που είναι βιώσιμα, διατηρούμε τις δεξιότητες μέσα από περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και προσελκύουμε επενδύσεις από έξω στις αγροτικές περιοχές διότι ε, ο κόσμος θέλει να ζει σε περιοχές που είναι δυναμικές και ελκυστικέ. Και είναι δύσκολο να ε, ποσοτικοποιήσουμε την συμβολή μας στο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το επόμενο ερώτημα είναι ποια από τα μέτρα που υπάρχουν στην ΚΑΠ αυτή τη στιγμή συμβάλλουν στην ε, τοποθεσία των ε, δημοσίων αγαθών. Έχουμε τον πρώτο πυλώνα, 40 δις ε, ευρώ το χρόνο. Αν δούμε τις άμεσες ενισχύσεις σε συνδυασμό με την πολλαπλή συμμόρφωση, υπάρχει κάποια συνεισφορά στα δημόσια αγαθά, σε μερικές περιπτώσεις ε, μπορεί να είναι, μην είναι και ο πρωτογενής στόχος. Στο πρώτο πυλώνα έχουμε τα πιο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα μέτρα στο άρθρο 68. Στον δεύτερο πυλώνα με στοχοθετημένα μέτρα, βλέπουμε μέτρα τα οποία είναι σχεδιασμένα να ε, δεσμεύσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ε, δημόσια αγαθά, ζωτικότητα της υπαίθρου, εδώ περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις για επενδύσεις, επίσης επιμόρφωση, ε, μεταφορά γνώσεων, ε, δημιουργία δυνατοτήτων. Αλλά δεν ανταποκρινόμαστε στους στόχους της φυσικοποικιλότητας, των κλιματικών αλλαγών και ενό επίπεδου συντήρησης των εδαφών. Δεν ανταποκρινόμαστε στους στόχους ε, των υδάτων. Και εδώ δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Άρα, αν θέλουμε να δούμε προς το μέλλον τι μέτρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στην κάποια για το σκοπό αυτό, κάποιες απλές αρχές, πρώτα απ' όλα χρειάζονται σαφείς στόχοι. Πρέπει, το πιο σημαντικό, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλα κίνητρα για τους αγρότες για να παρέχουν αυτά τα αγαθά και αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που είναι καλά σχεδιασμένα, εστιασμένα με συγκεκριμένο τρόπο, να μην είναι ασαφή και αναποτελεσματικά. Θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό τρόπο υλοποίηση και στοχοθέτηση. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση στην ΚΑΠ και έχουμε κάποιες, κάνει μελέτε που δείχνουν ότι πρέπει να δαπανείται ένα μεγάλο ποσό για να αποδίδονται τα δημοσία αγαθά στην Γεωργία. Δεν είναι, ε, μιλάμε για μικρά ποσά, είναι ένα μεγάλο στοιχείο, της, μεγάλο μέρο της ΚΑΠ, αν χρησιμοποιούμε τα δημόσια αγαθά ως κεντρικό στόχο. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, θα πρέπει να έχουμε σύμβουλες και κατάρτιση. Ε, οι γεωργοί χρειάζονται βοήθεια στο να προσαρμοστούν στην αποτελεσματική παραγωγή δημοσίων αγαθών. Πρέπει να υπάρχει διοικητική δυνατότητα και εμπειρογνωμοσύνη, καλή διαθεσιμότητα δεδομένων, παρακολούθηση και έλεγχος και πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση ανάμεσα στις ρυθμίσεις και στα κίνητρα. Και εδώ έρχομαστε σε ένα ερώτημα που η Επιτροπή έχει συζητήσει με την έκθεση του κυρίου Ντές σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα εδώ. Έχουμε μέτρα τα οποία είναι απλά, εύκολα και ευκατανόητα από τους ε, αγρότες και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα. Υπάρχουν άλλα μέτρα που είναι αποδοτικά, αποτελεσματικά, με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, που είναι ευαίσθητα σε θέματα παραγωγής, περιβάλλοντος. Δεν μπορείς να έχεις ένα που να ταιριάζει σε όλα, σε όλα τα περιβαλλοντικά προϊόντα. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν ανησυχούμε, αν αυξηθεί ε, ο αντίκτυπος, αν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα τοπία στην Ευρώπη δεν μπορούμε να έχουμε μια απλή συνταγή που να εφαρμόζεται σε κάθε κατάσταση και παντού. Άρα, έχουμε ένα δίλημα. Αφενός, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στοχευμένα μέτρα με κίνητρα που να παρακολουθούνται αποδοτικά, με feedback και ανατροφοδότηση. Γι' αυτό χρειάζεται προγραμματισμός και διοικητική εξειδίκευση, όχι σε επίπεδο εκμετάλλευσης, αλλά οι εθνικές και τοπικές δικής πρέπει να ξέρουν αυτά τα θέματα και πρέπει να υπάρχουν σωστά δεδομένα. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά του δεύτερου πυλώνα. Μπορούμε να δούμε ότι αφενός πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ε, όσο μπορούμε με μέτρα που να είναι απλά, σχετικά απλά, μπορεί να είναι πανευρωπαϊκά και σε άλλα μέτρα πρέπει να πούμε εντάξει, μπορεί να μην έχουμε δημόσια αγαθά, αν δεν έχουμε μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση και να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση της πυλώνα 2 περισσότερο. Στην πελέτη μας προτείναμε να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε κάπως τα μέσα και τα εργαλεία που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε στην ΚΑΠ σε τρία επίπεδα, σε τρία μπλοκ. Το πρώτο είναι τα σχετικά εύκολα που θα εφαρμόζονται σε ενδυνάμει όλες τις εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης και ε, έχει κάποιο όφελος κάθε εκμετάλλευση. Οι προτάσεις εδώ που θα τις ε, ε, αναπτύξουμε στην τελική έκθεση έχουμε τις οικολογικές αγραναπαύσεις, η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, των εκμεταλλεύσεων και απλά σχέδια έτσι ώστε οι αγρότες να σκεφτούν πώς μπορούν να διαχειριστούν τα εδάφη τους, πώς μπορούν να ε, διαχειριστούν τα ζωτούχα και τον άνθρακα στις εκμεταλλεύσεις. Τα εκμεταλλεύσεις που το κάνουν είναι ε, σημαντικό γιατί πάνε προς την κατεύθυνση της ε, παράδοσης καλών δημοσίων αγαθών. Μπορούν να προσαρτηθούν αυτά σε άμεσες ενισχύσεις πυλώνα 1. Ένα δεύτερο μπλοκ ε, μέτρων για τα δημόσια αγαθά είναι αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλες ε, ευρείες περιοχές της Ευρώπης η προστασία των ε, περιοχών των βοσκοτόπων, η διατήρηση της βιολογικής παραγωγής, Εκεί θα πρέπει να ποικίλει η στήριξη ανάλογα με τον πληθυσμό ε, το, την πυκνότητα πληθυσμού, ε, κτηνοτροφικού πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων. Αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι στον πυλώνα 1 ή σε προσέγγιση πυλώνα 2. Και τέλος, πολύ ε, στοχευμένα μέτρα τοπικά όπως επενδυτική βοήθεια, κατάρτιση. Αυτά είναι θελοντικά είναι ε, της προσέγγισης του πυλώνα 2 περισσότερο. Αυτή είναι μια μακροεικόνα της ΚΑΠ για το θέμα πυλώνα, μέτρων πυλώνα 1 και 2, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα και θα τα δω εντάχει. Θα πρέπει να έχουμε δημόσια αγαθά, στη που να υλοποιούνται παντού. Πολλά μέτρα δεν ε, υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά και το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να ενοποιήσουμε τα πρότυπα ΓΚΑΕΚ e και να διευκρινίσουμε την διάκριση ανάμεσα στην πολλαπλή συμμόρφωση και τις πληρωμές για τα πράσινα μέτρα του πυλώνα 1. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος ευκαιρίας σε αγροπεριβαλλοντικές πληρωμές. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να γράφονται οι γεωργοί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος προσδιορισμός κονδυλίων στον πυλώνα 2, έτσι ώστε να έχουν τα κίνητρα οι ε, αγρότες να δαπανίσουν ε, κονδύλια σε δημόσια αγαθά του πυλώνα 2. Αυτή είναι μια δίκαιη και συνεχτική εφαρμογή αυτού του κανόνα και τέλος θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξη της αγροτικής ζωτικότητας που πρέπει να είναι εντός πυλώνα 2 και τέλος δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα θέματα δημοσίων αγαθών. Είναι δύσκολο να δούμε σύστημα απόδοσης της ΚΑΠ που θα εφαρμοζόταν σε μικρές εκμεταλλεύσεις. Είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες, πολύ γραφειοκρατικές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα απλουστευμένο σύστημα για μικρές εκμεταλλεύσεις. Εδώ έχω τρία μπλοκ, τρία κοτιά. Για να σας δώσω μια ιδέα των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή για το πρασίνισμα του πυλώνα 1, τι πρέπει να παραμείνει, τι πρέπει να πάει στην προσέγγιση πυλώνα 2. Κάποιες από τις προτάσεις μας είναι κάπου στη μέση, όπου λέμε διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, ε, περιβαλλοντικές περιοχές προτεραιότητας άλλα μέτρα όπως η διατήρηση των βιολογικών καλλιεργιών μπορούν να πάνε είτε στον πυλώνα 1 είτε στον πυλώνα 2. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει, ε, υπάρχουν συμβουλές και δημιουργία δυνατοτήτων για τους γεωργούς. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα αναφοράς μέσα από την Επιτροπή. Ε, ε, θα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι που να εφαρμόζονται. Τώρα δύο άλλα θέματα πρωτού τελειώσω. Πρώτον, το πολύ δύσκολο θέμα της συγχρηματοδότησης και μια από τις ηρωνίες της ΚΑΠ είναι ότι εκεί που έχουμε πολιτικές με πολύ υψηλά ε, στοιχείο δημοσίων αγαθών όπως μέτρα δεύτερου πυλώνα έχουμε χαμηλότερη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό είναι κάπως περίεργο. Είναι γι' αυτό που δώσαμε έμφαση στο πρασίνισμα του πυλώνα 1. Πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν να δαπανίσουν μεγάλα ποσά σε μέτρα του πυλώνα 2, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση και αυτό είναι ε, ένα σημείο που ακριβώς όπως λειτουργεί η συγχρηματοδότηση. Δεν πρέπει αυτό να οθεί την όλη ανταπόκριση το δίλημα της πολιτικής. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή πολιτική για το σωστό, στοχό, ε, σωστό σκοπό. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί και να πούμε ότι τελικά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση ε, ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό δημοσίου συμφέροντος. Και τέλος δεν μπορείς να έχεις απόδοση σε όλα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά ή τα κοινωνικά δημόσια αγαθά μέσα από την ΚΑΠ χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα. Μη ΚΑΠ, για παράδειγμα στήριξη ή παρέμβαση μέσα από άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, τα διαρθρωτικά ταμεία, LIFE κλπ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι εμπλοκής ε, της αγοράς. Επίσης ε, ιδιωτικό ενδιαφέρον όπως ε, εταιρείε υδάτων που χρηματοδοτούν τους αγρότες. Είναι σε μικρή κλίμακα ακόμα και μακροχρόνια θα πρέπει να δώσουμε περαιτέρω σημασία σε αυτό. Επίσης, χρειαζόμαστε σίγουρα καινοτομία, ανάπτυξη τεχνολογική, έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό αφορά και παραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Εδώ πρέπει να γίνει επένδυση στον τεχνολογικό τομέα. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι αυτά που συμβαίνουν στη Γεωργία οθούνται από πολιτικές ενεργειακές εκτός της ΚΑΠ και αν θέλουμε μια αηφόρο και ε, χρήσιμη ΚΑΠ ε, θα πρέπει να ε, την συνδυάσουμε με αυτές τις άλλες, αυτά τα άλλα κίνητρα. Επίσης, ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Το, το, σημαντικό μήνυμα εδώ είναι ότι βλέπουμε ότι είναι πολύ δυνατόν να αναπτυχθούν εφικτά μέτρα εντός της ΚΑΠ ε, για να παρέχουμε δημόσια αγαθά. Αυτά δεν θα είναι πάντα συμβατά με την ε, απλοϊκή προσέγγιση. Για άλλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερη προσοχή, να χρειαστεί περισσότερη προσοχή. Προσβλέπουμε στα σχόλιά σας, στις αντιδράσεις σας, προτού εκδώσουμε την τελική μας έκθεση. Σας ευχαριστώ. Mr. give the floor. Κύριε Ντέσ, να σας δώσω το λόγο, παρακαλώ. Κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Και πολύ λυπάμαι που πολλοί συνάδελφοι δεν είναι πλέον στην αίθουσα. Που έχουν εντελώ αντίθετη άποψη σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τον νέο προσανατολισμό της γεωργικής πολιτικής και στην ομάδα μου και σε άλλες ομάδες. Καλό είναι να ακούμε τέτοιες παρουσιάσεις και βλέπω ότι συμφωνείτε με τις σκέψεις τις οποίες χρησιμοποίησα για την έκθεση. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένα κάποιο πρόβλημα κατανόησης, αλλά ανακύπτει και πάλι το ερώτημα πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια σύγχυση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Μια εικόνα με ενόχλησε κάπως, όπως στη μέση ήταν ο πιο παχής πυλώνας. Τι είχατε υπόψη σας, γιατί δηλαδή ήταν τόσο πιο μεγάλος ο πυλώνας ο μεσαίος μεταξύ πρώτου και τρίτου. Νομίζω ότι εδώ είναι απαραίτητο να το συζητήσουμε. Mr. Agnew. Κύριε Σαγνιού. Ναι. Κάποιες ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Η μία είναι μάλλον προβλέψιμη. Λέτε ότι οι αγρότες θα παρέχουν ένα κοινό αγαθό αν μειώσουν τις εκπομπές τους. Να κοιτάξουμε το μεθάνιο. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μεθανίου στη γεωργία, θα πρέπει να περιοριστούν να μειωθούν τα αποθέματα, τα κοπάδια. Άρα θα πρέπει να περιοριστούν δηλαδή τα αμερικαστικά. Ο μοναδικός, ε, είναι η μοναδική λογική που βλέπω στο επιχειρημα, στην επιχειρηματολογία ε, σας. Η άλλη πρόταση που κάνετε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι βιολογικοί αγρότες θα παραμείνουν βιολογικοί. Ο τομέας αυτός θα πρέπει να ακολουθήσει τους καταναλωτές. Ο κόσμος που πάει στα μαγαζιά και ζητάει βιολογικά προϊόντα είναι αυτό καθορίζει πόσα εκτάρια, τι επιφάνεια καλλιεργείται βιολογικά. Αν εμεί βγούμε και πούμε ότι ε, θέλουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό εκταρίων να καλλιεργούνται με βιολογικά προϊόντα, αυτό θα προκαλέσει κατάρρευση των τιμών. Και θα μειωθεί τελικά ο καταναλωτή. Ούτε νομίζω ότι θα ωφελήσουμε τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων επιβάλλοντας τέτοιους ε, περιορισμούς. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και για την παρουσίαση τέργεζα πραγματικά και με την προηγούμενη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την υπόδειξη αυτή. Μας παρουσιάστηκαν και οι αντιφάσεις. Προσπαθούμε στην αγροτική μεταρρύθμιση να δούμε και αυτή τη διάθεση κοινών αγαθών και να δώσουμε και ένα πράσινο χαρακτήρα, μια πράσινη όψη σε αυτό στη μελέτη βρήκα και τρία βασικά επιχειρήματα που μας απασχολούν και τα οποία λένε ότι εντάξει τα αναγνωρίζουμε, θέλουμε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Γεωργία να παράγουν καταρχάς και σε πρώτο, σε πρώτο βαθμό τρόφιμα. Υπάρχουν όμως τρία προβλήματα τα οποία ανέφερε εν μέρη και η μελέτη. Το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής. Στην ε, νέα αγροτική μεταρρύθμιση αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη τον πράσινο χαρακτήρα, θέλουμε να δαπανίσουμε χρήματα, δεν θέλουμε όμως ο αγρότης να βρεθεί με ένα νέο τελείως ε, μηχανισμό ελέγχου. Είπατε πολύ ορθά ότι αν θέλουμε να εισάγουμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και ένα μηχανισμό αναφοράς και ελέγχου. Αλλά εμείς έχουμε ήδη δύο τέτοιους μηχανισμούς. Ένα με την πολλαπλή συμμόρφωση τον οποίο ε, τον γνωρίζουν πλέον οι γεωργοί και έναν μηχανισμό ελέγχου στο δεύτερο πυλώνα σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Έρωτα λοιπόν αν σωστά κατάλαβα ή μήπως δεν κατάλαβα σωστά αυτός ο μηχανισμός ε, αναφοράς και ελέγχου για το πρασίνισμα των ε, αγαθών. Πού θέλετε να μπει. Κατά δεύτερον, διαπιστώνεται και δικαίως ότι το, βασικά, το βασικό πρόβλημα είναι ότι στο δεύτερο πυλώνα κάποια κράτη-μέλη δεν θα έχουν χρήματα για την συγχρηματοδότηση. Άρα, λέτε να παραμείνουμε στον πρώτο πυλώνα όπου δεν χρειάζεται συγχρηματοδότηση. Ρωτώ, μπορείτε να φανταστείτε να συμπεριληφθούν τα προγράμματα αυτά στο δεύτερο πυλώνα χωρίς συγχρηματοδότηση όμως θεωρείτε ότι θα αποτελούσε και αυτό μια ενδεχόμενη λύση. Και τρίτη ερώτηση που κατά πάσα πιθανότητα μας απασχολεί πιο πολύ ως ε, αγροτικού, πολιτικού συντομέα της γεωργίας και λιγότερο σε ό,τι αφορά την μελέτη. Υπάρχουν ε, μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για όλους. Και κατά δεύτερον υπάρχουν μέτρα που είναι πολύ ειδικά είναι σημαντικό λοιπόν, μάλλον η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική, γιατί τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και φοβόμαστε, και θα επανέλθω στο σημείο αυτό στην έκθεση DES, φοβόμαστε, μάλλον αυτό που δεν επιτρέπεται να συμβεί είναι το εξή. Με τα εφιστάμενα καινούργια προγράμματα, με τα νέα μέτρα πρασινίσματος, να καταστραφούν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα. Δεν είμαστε σοβαροί όταν λέμε ότι ο αγρότης θα πρέπει να λάβει μέτρα για το πρασίνισμα, θα πάρει 60 ευρώ ανακτάριο και κατά δεύτερον, αλλά κατά δεύτερον στο στον τομέα του δεύτερου πυλώνα θα του αφαιρεθούν προγράμματα περιβαλλοντικά. Αυτό δεν έχει νόημα. Και τελικά θα χάσει. Να δούμε λοιπόν να υπάρχει μια κάποια λογική μεταξύ των προγραμμάτων για το πρασίνισμα της οικονομίας και των ήδη φυστάμενων προγραμμάτων. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας πήρα σχεδόν τη θέση. Ευτυχώς που γυρίσατε. Ευχαριστώ πολύ για τους συντάκτες ε, της έκθεσης. Ε, θα ήθελα να σταθώ στις διαφάνειες 7 και 8 διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στην 7 λέμε ότι οι άμεσες ε, ενισχύσεις με την διασταυρούμενη συμμόρφωση θα συνεισφέρουν στα δημόσια αγαθά δεν είναι ο σκοπός τους αυτός. Ε, έχει σημασία το γεγονός ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το παρόν σύστημα έχει αποτελέσματα με τα δημόσια αγαθά. Αν θέλουμε λοιπόν να εμβαθύνουμε στο επίπεδο των ε, δημοσίων αγαθών που μας παρέχει η Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής του κλίματος, της βιοπικιλότητας, ε, το έδαφος και το είδωρ, μήπως θα έπρεπε να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατανομής στον προπολογισμό. Τώρα, Στη διαφάνεια παριθμών 8 στην παρουσίαση αναφέρεστε σε επαρκείς ε, πόρους από τον προπολογισμό. Ίσως θα έπρεπε να μας δώσετε κάποια περαιτέρω στοιχείο. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση του προπολογισμού είναι πολύ δύσκολη. Πείτε μας τι εννοείτε. Το επόμενο στοιχείο που θέλω να αναφέρω αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων. Θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο περαιτέρω το θέμα αυτό Λέτε ότι στη μεταρρύθμιση για την ΚΑΠ θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης για τους γεωργιούς. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πλέον δημόσια υποστήριξη για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, ίσως και για την έρευνα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα θέλαμε λοιπόν τα σχόλιά σας επ' αυτού. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να δαπανούμε πολλά κονδύλια για να παραδίδουμε δημόσια αγαθά. Και πάλι θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό διότι εγώ διαπίστωσα και νομίζω ότι και ο Επίτροπος Ποτότσνικ συμφωνεί με αυτή την παρατήρηση ότι οι... όσοι ασχολούνται με τη γεωργία θεωρούν ότι οι γεωργοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι να μας δώσουν στοιχεία για το περιβάλλον γιατί θα μας το κάνουν φθηνά. Οποιοςδήποτε άλλος θα χρησιμοποιήσει πολύ πιο διαπανερό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε στοιχεία. Πώς μπορούμε να έχουμε αξία από την ΚΑΠ. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε αυτό. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι θα ήθελα να είχα αυτή τη μελέτη πριν από δύο χρόνια και όχι τώρα, διότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο στι διαπραγματεύσει. Επομένω, θα ήταν πολύ χρήσιμο να την είχαμε στο παρελθόν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαγκίνα και να δώσω τώρα το λόγο στου συγητέ. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο, ο Κοράντο, παρακαλώ. Εγώ θα αναφερθώ σε τρία πράγματα και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει ο Ντέιβιτ. Το πρώτο αφορά τις εκπομπές μεθανίου. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. διότι το μεθάνιο ως παραπροϊόν ε, της κτηνοτροφίας δεν έχει ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για την αλλαγή του κλίματος, που έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στο διοξίδιο του άνθρακα και όχι τόσο στο μεθάνιο. Θεωρώ ότι εδώ πριν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση, μπορεί να μην έχουμε και πολλά στοιχεία, διότι είναι περίπλοκο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα από τώρα ήδη, διότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Μέχρι τούδε επικεντρωθήκαμε τα βιοκαύσιμα, τα οποία αποτελούν επιπλέον εισόδημα για τους ε, γεωργούς, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Ίσως όμως αύριο να πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε κίνητρα για τους γεωργούς για να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη πολιτική ζευγαρώματος των ζώων που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το εισόδημα επιπλέον για τους ε, γεωργούς, αλλά θα ασχολείται αποτελεσματικά με τα απόβλητα και την ε, σωστή τους διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη πολιτική, διότι όταν θα αρχίσουμε να συζητάμε για τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά κίνητρα και την ε, τιμολόγηση που θα ισχύει για την ενέργεια και για άλλα στοιχεία, μέτρα υποστήριξης της αγοράς όπως για παράδειγμα πράσινα πιστοποιητικά, και άλλα ρυθμιστικά στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητο ε, στοιχείο της ΚΑΠ, αλλά άλλα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να επιλύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του βιολογικού. Είναι σωστό ότι σε κάποιες ε, περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν υπάρχει πλέον βιολογική παραγωγή. Θυμάμαι ότι κάποιος κάποτε είπε ότι η βιολογική γεωργική παραγωγή στη Γερμανία θα πρέπει να φτάσει στο 20%. αυτό ήταν ανεύθυνο. Ανακοινώνεται μια πολιτική της κυβέρνησης ε, προς τους παραγωγούς με στόχο κατά 20% και ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη παραγωγή βιολογικών προϊόντων ενώ δεν υπάρχει ζήτηση. Και αυτό είναι λανθασμένο διότι η ζήτηση είναι βασική για τον παραγωγό. Αν δεν υπάρχει πλέον αγορά για ένα προϊόν ή δεν είναι επαρκή, δεν αναπτύσσεται ε, κατάλληλα, η παραγωγή του πάει στα σκουπίδια και αυτό φυσικά αποθαρρύνει την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενώ κανονικά θα έπρεπε να την ευνοούμε. Εδώ είναι θέμα πολιτικής μας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες ότι πρόκειται για σημαντικό στοιχείο. Μπορεί να μιλήσουμε και για χρηματοοικονομικά κίνητρα. Καλώ. Χωρίς αυτά ε, οι γεωργοί δεν θα κάνουν είτε είναι υποχρεωτικό είτε όχι αυτό που απαιτείται. Εάν δεν υπάρχουν κίνητρα. Εγώ δεν βλέπω κίνητρα προ το παρόν, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ξυπνήσουμε. Υπάρχει όμω και το θέμα των συμβουλών δεν μπορεί να περιμένουμε από τους γεωργούς να προσαρμόσουν τον τρόπο παραγωγής τους, να κάνουν νέα πράγματα και να παράγουν δημόσια αγαθά χωρίς να γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Ο Γεωργός δεν θέλει να κινδυνεύσει να χάσει τη δουλειά του και να χάσει τα εισοδήματα που έχει. Επομένως χρειάζεται ούτως ή άλλως ε, συμβουλή και όχι εγγύηση, αλλά μια ενθάρρυνση που θα του λέει ότι αν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής του δεν θα έχει ε, οικονομικές ε, ζημίες. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι όπως είπε ο Ντέιβιντ, εάν κάποιος προωθεί δημόσια αγαθά και πιέζουμε αυτή την παραγωγή, θα δημιουργηθούν πολύ περίπλοκη κατάσταση. Μπορεί να το αναμάστε όπως θέλετε, να χρησιμοποιείτε τον όρο απρούστευση κάθε πέντε λεπτά, αλλά αν γίνουν έτσι τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα. Ας το δεχτούμε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε την κατάσταση. Διότι παρόλο που θα είναι πιο περίπλοκο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι για να το απλουστεύσουμε ως αντιστάθμισμα. Και εδώ, και το συζητούσαμε αυτό σήμερα το πρωί, έγκυται και το θέμα της συμβουλευτικής υπηρεσίας, της παρακολούθησης και ταυτόχρονα και της εποπτείας και του ελέγχου. Αυτή τη στιγμή ο Γιωργός έχει διάφορες επισκέψεις για το τάδε, το δίνα και το άλλο το τρίτο. Εάν λοιπόν δεν απλουστεύσουμε τα πράγματα, απλώς θα τον ενοχλούν διάφοροι και θα χάνει την ώρα του για γραφειοκρατία. μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο ίσως θα το επικρίνουν, αλλά θα είναι λίγο πρωτότυπο και θα έχει μια χρησιμότητα για τον Γιώργο. Να συνδυάσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα σε μία επίσκεψη και να υπάρχει ταυτόχρονα και συμβουλευτική υπηρεσία. Εάν δεν αρέσουν ε, στο Γιώργο πολλοί επισκέψεις ε, για, ε, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, όλα θα του αρέσουν οι συμβουλές. Εάν κάποιος λοιπόν παρακολουθεί τα πράγματα και διαπιστώσει ότι κάτι είναι λανθασμένο ή κάποιος ελέγχει και διαπιστώνει ότι κάτι έχει πάει στραβά, ο μόνος λόγος, ο τρόπος θα ήταν να το τιμωρήσουμε. Αλλά έτσι δεν λύνουμε το πρόβλημα. Ιδίω στη στάδια της παρακολούθησης θα μπορούσε κάποιος εκ των προτέρων να κάνει πράγματα ώστε να μην πάει στράφη ο έλεγχος. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν δοθούν κίνητρα στον Γεωργό και προσθέσουμε και τις συμβουλές. Γιατί να μην γίνονται κοινέ επισκέψει, όπου θα υπάρχει το συμβουλευτικό κομμάτι, κάποιο διαφορετικό κλάδο. Δεν έχει σημασία ποιο θα είναι, αλλά θα υπάρχει ένα σύμβουλο, θα υπάρχει αυτό που κάνει την παρακολούθηση και θα υπάρχει και αυτό που κάνει τον έλεγχο. Και θα είναι όλοι εκεί και κατά κάποιον τρόπο θα ακούν ο ένα και από τον άλλον ποια είναι τα προβλήματα. Μπορεί ο σύμβουλο να πει σε αυτού που ελέγχουν και παρακολουθούν ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρί το άλλο, χωρί τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλιώ δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Και τότε αυτοί που κάνουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο μπορεί να μάθουν και κάτι από τον ε, σύμβουλο για τρόπου επίλυση προβλημάτων. Και ο Γεωργό από καιρού ει καιρών θα πρέπει να υποστεί μόνο μια επίσκεψη που θα εξετάζει όλε τι πτυχές. Τον πρώτο πυλώνα, το δεύτερο πυλώνα, τα συμβουλευτικά θέματα, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Εάν δεν δαπανίσουμε περισσότερα κονδύλια για τις συμβουλές και όχι μόνο στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι ό,τι συζητάμε για τα δημόσια αγαθά δυστυχώς δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κοράντο. Θέλει και ο Ντέιβιτ το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω εν συντομία σε ορισμένα από τα άλλα ερωτήματα που δεν απέντησε ο Κοράντο. Ένα, είναι το θέμα του τρίτου πυλώνα. Ο κύριος Ντες το ανέφερε. Δεν προτείνουμε ένα τρίτο πυλώνα. Λυπάμαι αν δεν έγινε σαφές. Αυτό που κάναμε στο σχεδιάγραμμα είναι βάλαμε ένα κουτί με κάποια μέτρα δημοσίων αγαθών που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προς ποια κατεύθυνση θα ε, κατευθυνθούν. Κάποια μπορεί εν δυνάμει να μπουν στο πυλώνα 1, άλλα στο πυλώνα 2. Αν διαβάσετε την πρόταση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή, έχουν δώσει μια πολύ ευρία περιγραφή με κάποια πιθανά παραδείγματα. Αυτό που λείπει είναι συγκεκριμένες προτάσεις ποια εντάσσονται σε ποιον πυλώνα και πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση λέγοντας, αν σκεφτούμε με συστηματικό τρόπο το, τα μέτρα πρασινίσματος, κάποια είναι αρκετά ε, απλά για τον πυλώνα 1, αλλά όχι. Άρα ε, μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά τα μέτρα δημοσίων αγαθών στο κατάλληλο Χρειάζεται όμως προσοχή. Δεν είναι μόνο πολιτικό θέμα, είναι και τεχνικό θέμα, διότι κάποια μέτρα θα πρέπει να παραδοθούν μέσα από ε, κάποιες διοικητικές δομές. Αν, ε, και υπάρχει και το, η πολιτική διάσταση φυσικά. Ένα, ένα δυο άλλα θέματα είναι η παρακολούθηση, λέμε ότι αν τα μέτρα είναι πιο στοχευμένα θα πρέπει να παρακολουθούνται. Η παρακολούθηση στο δεύτερο πυλώνα πετυχαίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ καλύτερο από την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε πιο εξελιγμένη παρακολούθηση εκεί. Αν θέλουμε δημόσια αγαθά στον πυλώνα 1 θα πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι επίπτωση. Έχουμε στοχευμένα ε, μέτρα, θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της Στο θέμα της συγχρηματοδότησης, το πυλώνα 2 υπάρχει μεγάλος διάλογος. Από θεωρητικής άποψης είναι ευκταίο να υπάρχουν πολιτικές ε, που να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει πρακτικό θέμα. Αν ε, παράγονται σε τοπικό επίπεδο μπορεί να γίνει ε, αποτελεσματικά. Χρειάζεται να συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη με τα κονδυλιά τους. Αυτό είναι το σοβαρό επιχείρημα κατά της χρηματοδότησης στον πυλώνα 2 κατά την άποψη. Μήπως υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ανάμεσα στον πυλώνα 1 και πυλώνα 2. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή διότι ο καθένας συζητάει για μέτρα τα οποία μπορούν να πάνε ή στον ένα ή στον άλλο πυλώνα. Ε, στον δεύτερο πυλώνα χρειάζονται πιο στοχευμένα μέτρα. Αλλά υπάρχουν κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να μπουν και στον πυλώνα 1. Θα πρέπει όμως να τα περιγράψουμε σύμφωνα με τον στόχο τους και τις τεχνικές δυνατότητές τους, αν ε, μπορούν να ενταχθούν σε μία προγραμματική περίοδο και χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν για θέματα όπως είναι η αξιολόγησή του σε ένα χρόνο, αν ε, πρέπει να πληρωθεί ο αγρότης εκείνο το χρόνο ή τον επόμενο χρόνο. Πρέπει να έχουμε δεσμεύσεις πολιετής ή ενός έτους. Αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν είναι πολιτικής φύσεως θέματα, αλλά θα πρέπει να είναι διαφανή και αν το Κοινοβούλιο θα μπει σε μια λεπτομερή γνωμοδότηση, θα πρέπει να τα δείτε και αυτά λεπτομερώς. Στο θέμα του προεπολογισμού, πόσα χρήματα χρειαζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες μελέτες στην Ευρώπη και έχουμε εκπονήσει και μία που δείχνουν ότι αν θέλουμε να αποδίδουμε και να παραδίδουμε όλους τους στόχους αποτελεσματικά και πλήρως και απέχουμε πολύ από αυτό το στόχο, θα μπορούσαμε να δαπάνουμε αν χρησιμοποιούσαμε θελοντικά σχέδια, 30 δις ευρώ το χρόνο κάνοντας αυτά, ίσως και περισσότερα. Άρα δεν συζητάμε εδώ για μεγάλες περικοπές της ΚΑΠ για την παράδοση αυτών των δημοσίων αγαθών. Μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος της ΚΑΠ που θα αφορά και άλλα θέματα εκτός από δημοσία αγαθά. Κάποιοι έχουν την ασφαλμένη ιδέα ότι αν τα ε, είναι φτηνή κάπου με τα δημόσια αγαθά. Όχι, αν θέλουμε να θέσουμε ψηλά πρότυπα. Εξαρτάται πόσο ψηλά είναι τα πρότυπα που θέλουμε να θέσουμε. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που ήθελα να απαντήσω. Κοράτο, θες να προσθέσεις και εσύ κάτι. Ναι, ναι. Θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα για τους πυλώνες. Νομίζω ότι τα δημόσια αγαθά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμπεριλαμβάνονται και στους δύο πυλώνες. Για τον απλό λόγο ότι εάν ε, τα έχουμε μόνο στο δεύτερο πυλώνα, εκεί έχουμε μόνο 13 δις. Δεν θα μας επιτρέπεται να κάνουμε αρκετά. Αφετέρου, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταβίβαση κονδυλίων από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2, διότι αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα εξ αρχής. Το ένα είναι ότι οι γεωργοί θα νιώσουν αυτομάτως την, απόλυτα, την απώλεια, διότι ο πυλώνας 2 δεν πηγαίνει απευθείας ε, στους γεωργούς. Και από την άλλη μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα με την δημοσιονομική αρχή. Θα μας πει η δημοσιονομική αρχή ότι μειώνεται τον πυλώνα 1, άρα να δώσουμε χρήματα πίσω στα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πάντα ελοχεύει ένα κίνδυνο όταν προσπαθούμε να μεταφέρουμε κονδύλιο. Από την άλλη βέβαια μπορούμε να έχουμε τις αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα ε, για τα δημόσια αγαθά. Αυτό έχει σχέση με το τι κάνουμε στον πρώτο πυλώνα και τι κάνουμε στο δεύτερο πυλώνα. Αν έχουμε καλές περιβαλλοντικές πλακτικές ε, στον πρώτο πυλώνα με τη διαμορφούμενη συμμόρφωση, τη διασταυρούμενη συμμόρφωση και τα όλα όσα σκεφτόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αν α, όμως η Επιτροπή πει ότι τα περιβαλλοντικά και γεωργικά μέτρα θα είναι εν μέρη στον πρώτο πυλώνα και εν μέρη στον δεύτερο πυλώνα, καλή τύχη να δω πώς θα τα διαχειριστούμε αυτά. Πέραν από τον προπολογισμό όμω, υπάρχει και αυτό που είπε ο Ντέιβιτ. Ούτω ή άλλω δεν επαρκεί ο προπολογισμό για να κάνουμε όσα απαιτούνται για τα δημόσια αγαθά. Ούτω ή άλλω δεν μα επαρκεί. Επομένω, Εάν τα δημόσια οικονομικά δεν επαρκούν για να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα για τους γεωργούς και τότε η προσέγγισή μας δεν θα έχει αποτέλεσμα. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχουν λύσεις που θα βασίζονται στην αγορά για να δίνονται ωφέλη για τις υπηρεσίες για τα οικοσυστήματα ε, μαζί με την καλή διαχείριση, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τα δημόσια αγαθά. Και υπάρχουν λύσεις. Το ένα είναι το Habitat Banking που αναφέρθηκε. Υπάρχουν αρκετές ε, τράπεζες ε, φυσικών οικοτόπων και κατά κάποιο τρόπο έχουν αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν λοιπόν να μας ε, παράσχουν πολύ σημαντικά ποσά χρημάτων Υποχρεώνοντα όσου εκμεταλλεύονται και αναπτύσσουν τη γη να πληρώνουν πιστώσει διότι ζημιώνουν το περιβάλλον και αυτά τα κονδύλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μακροπρόθεσμε επενδύσει για του γεωργού. Και από πλευρά υδάτων δεν νομίζω ότι μπορούμε απλώς να επιβάλλουμε κανονισμό στους γεωργούς για να τους ακολουθήσουν με επιπλέον κόστος χωρίς να υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση, γιατί δεν θα υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση. Και εκεί υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγματα συμφωνιών μεταξύ εταιριών υδάτων, ακόμα και ιδιωτικών εταιριών ε, ε, νερού όπως η Βιτέλ και γεωργών που λένε το εξής. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό ως γεωργός για να διατηρήσεις τα ύδατα καθαρά και αν το κάνεις αυτό εγώ θα σου δώσω χρήματα γιατί αν μου καταστρέψει το νερό μου η Βιτέλ θα χρεοκοπήσει γιατί κανείς δεν θα αγοράζει μολυσμένο νερό και οι εταιρείε υδάτων λένε ότι αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, θα πρέπει εγώ να κάνω καθαρισμό ύδατο και επομένω θα πληρώσω πολλά χρήματα. Προτιμώ να σου δώσω ένα τα μισά, να κερδίσει εσύ κάποια χρήματα για τη διατηρήση το νερό μου καθαρό, ακολουθεί την ε, οδηγία για τα ύδατα και ταυτόχρονα εγώ αποταμιώβω γιατί ε, ξοδεύω λιγότερα για, την αποταμίευση... για τον καθαρισμό του νερού. Συγγνώμη αν έχουμε ένα σύστημα, δεν αναφέρομαι στο σύστημα εμπορία εκπομπών που θα περιλαμβάνει και γεωργικά προϊόντα, αλλά πιο περιορισμένα πράγματα. Συμβάσει με εταιρείε υδάτων ή με εταιρείε ε, που παρέχουν ε, ε, νερό και τους γεωργούς και έτσι θα έχουμε λιγότερες δυσκολίες και θα πείσουμε πιο εύκολα τους γεωργούς να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε ειλικρινώ, λέει ο πρόεδρο, τον Ντέιβιτ Πάλκοβ και τον Κοράντο Πρίτσιο Μπύρολη. Μα έχουν δώσει πολλά ενάψματα για συζήτηση με, με τη μελέτη αυτή και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον Τάσο, τον Μπασκού, τον Μπόσαρτ και όλους τους ευρωβουλευτές και νομίζω ότι πλέον, επειδή δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διήμερη συνεδρία της Επιτροπής μας, η οποία ήταν πλουσιότατη. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 2 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι.